Oh, maybe they'll come. Ladies and gentlemen, good e- Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ, καθίστε. Ελπίζω να με ακούτε. Είμαι λίγο βραχνιασμένη, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σας καλησπερίζω λοιπόν όλους στην πρώτη αυτή συνάντηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας βλέπω καλά, περάσατε καλά, οπότε προχωράμε αμέσως να σας υπενθυμίσω ότι ε, αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνάντηση. σε επίπεδο διερμηνίας είναι διαθέσιμες συγκεκριμένες γλώσσες με βάση τις προτεραιότητες που έχουμε των μελών της ε, Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Ας ξεκινήσω με τα πρακτικά. Να σας υπενθυμίσω με την ημερήσια διάταξη, συγγνώμη, Υπήρξε μια συνάντηση στο τέλος της ε, προηγούμενης συνάντησής μας και αποφασίσαμε να ανταλλάξουμε τη σειρά ανάμεσα στο σημείο 6 ενημέρωση για την αποστολή της ΣΕΝΤΕ στην Ιταλία και γενικότερα στη Μεσόγειο. Η αποστολή αυτή έγινε μετά τις 15 Ιουλίου. και μετά θα συζητήσουμε την έκθεση, την ετήσια για την ΚΕΠΑ. Λοιπόν, θεωρώ ότι μια και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις γίνεται δεκτή η μερίσια διάταξη. Περνάω λοιπόν τώρα στα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. 21ης και 22ης Ιουνίου αν έχετε κάποια παρατήρηση μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Τη απουσία παρατηρήσεων θεωρούνται δεκτά τα πρακτικά. Όπως γνωρίζετε, σήμερα Έχουμε την συμπληρωματική εκλογή του τρίτου μέλους της υποεπιτροπής, του Προεδρείου της Υποεπιτροπής, δηλαδή του Αντιπροέδρου, ο κύριος Χάσελκαμπ, εξελέγει εν το μεταξύ που ήταν Αντιπρόεδρος, στην Κάτω Βουλή, μετά από τις τελευταίες εκλογές και γι' αυτό χειρεύει η, η θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Από ό,τι φαίνεται, μία υποψηφιότητα έχει κατατεθεί, η κυρία Μούντι, για τους σοσιαλιστές. Θα ήθελα να μου ανακοινώσετε αν υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μποστινάρου να μας παρουσιάσει την υποψηφιότητα της Κλέα Μούντι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εξ ονόματος των μελών της ομάδας μου και των συντονιστών μας, του συντονιστή μας του κ. Πάσκου, εμείς εμπιστευόμεθα και συνεπώς θα στηρίξουμε την κυρία Μούντι στην προσπάθειά της να γίνει μέλος του Προεδρείου της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Και γι' αυτό θα ήθελα παρακαλώ να βοηθήσετε να εκλεγεί ήδη από σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφε. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις παρακαλώ σχετικά με την υποψηφιότητα της κυρίας Μούντι. Θέλετε να γίνει μυστική ψηφοφορία. Νομίζω όμως ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά την κυρία Μούντι από τις δραστηριότητές της σε διάφορα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα. Και γι' αυτό με την άδειά σας, εφόσον συμφωνείτε, διαβοής παρακαλώ ή η αποδοχή της υποψηφιότητας Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Συνεπώς περνάμε απευθείας στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να συγχαρώ πρώτα την κυρία Μούντι Φυσικά και αυτή έχει τη δυνατότητα να έρθει στο Προεδρείο. Θα ζητήσω τώρα από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μας, τους προσκεκλημένους, να πάρουν τις θέσεις τους.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 Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, ο τίτλος του επόμενου θέματος είναι οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στον μετασοβιετικό χώρο. Mm. Ιδιαιτέρως στην Ουκρανία και την Μπελαρούς, Λευκορωσία στόχος αυτής της δημόσιας ακρόασης, γιατί είναι επαναλαμβάνω δημόσια, είναι να παρουσιαστούν οι περίπλοκες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή αυτή, ιδιαιτέρως λόγω πριν ε, της ε, διεξαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων Ζαπάντ 17 ανάμεσα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις, αυτά τα στρατιωτικά γυμνάσια περιλαμβάνουν πάρα πολύ υψηλό αριθμό στρατευμάτων που συμμετέχουν. Θα καλύψουν περίπου το σύνολο της περιοχής και υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τον σεβασμό της Διεθνούς Συμφωνίας για την παρακολούθηση της ασκήσεως Ζαπάντα. Η δημοκρατική κοινότης θεωρεί ότι οι στρατιωτικές αυτές ασκήσεις είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικές και ιδιαιτέρως επικίνδυνες. Λοιπόν, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τους εμπειρογνώμονες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε σωστά ενημερωμένοι για το σύνολο των προβλημάτων της περιοχής. Ας καλωσορίσω λοιπόν τον υποδιευθυντή της EEAS, τον κύριο Λιουκ Ντεβίνια, υπεύθυνο για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε επίσης ε, και έναν γνωστό εμπειρογνώμονα, πολύ γνωστό και εδώ στο Κοινοβούλιο, από γεγονότα τα οποία είχαν ε, οργανωθεί ακριβώς επανειλημμένα στο παρελθόν Θυμάμαι τις παρατηρήσεις τις οποίες είχε κάνει στην Ρήγα στα πλαίσια της ε, διακοινοβουλευτικής συνάντησης για την ΚΕΠΑ και θέματα ασφάλειας γενικά. Είχε οργανωθεί από τη Λετωνική Προεδρία. Επίσης έχουμε και τον κύριο James Share γνωστός εμπειρογνώμονας από το Think Tank Chatham House του Λονδίνου. Και έχουμε επίσης και τον κύριο Ράτς στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. και επίσης ένας επιπλέον πολύ γνωστός εμπειρογνώμων είναι η Άννα Μαρία Ντίνερ αναλύτρια στο Πολωνικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων. Χωρίς λοιπόν άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στους διακεκριμένους ομιλητές μας. Να πω επίσης ότι αυτή εδώ η δημόσια ακρόαση οργανώνεται σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ουκρανία, Λευκορωσία και Ρωσία. Κάποιοι από τους υπεύθυνους των αντιπροσωπιών αυτών είναι εδώ παρόντες. Καλώς λοιπόν κυρίες και κύριοι, δίνω το λόγο στον κύριο Ντεβίνια. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα αξιότιμη μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Με χαρά έρχομαι ενώπιον της Επιτροπής το θέμα είναι ευρύτατο όσο και σημαντικότατο όπως όλοι γνωρίζουμε. Η διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ήταν στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από την αρχή του. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έφερε επιπλέον ευθύνε για να δούμε τι θα γίνει με τις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια στα ανατολικά της Ήπειρου μας. Έχουμε μια ευρεία στρατηγική και πολιτική γειτονία που τα αντανακλούν όλα αυτά. Όπως είδαμε στην κρίση εντός και γύρω από την Ουκρανία, δυστυχώς ε, μη σεβασμός της ε, τάξης της Ευρωπαϊκής και της ασφάλειας που έχει να κάνει με το σεβασμό και ε, την προστασία των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών Καθώ επίσης και τι αρχές τη αυτοδιάθεση των λαών ε, που παραβιάζεται, ε, συνιστούν ε, προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προσέγγιση της σχετικά με την περιοχή, αλλά και όλη την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τελικά την ευημερία στην Ευρώπη, ο μόνος δρόμος είναι οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλοι ενιστούμε ένα καλύτερο μέλλον για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού μας όταν πρόκειται για την προώθηση της ασφάλειας στην άμεση γειτονία μας. Θα ήθελα καταρχάς να πω δύο λόγια για το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί τα ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας ανατολικά. Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε πρόσφατες εξελίξεις και τέλος ε, πώς ε, θα βοηθήσουμε ε, για να γεφυρωθούν τα χάσματα, να επανέλθει η συμφιλίωση και θα αναφερθώ στη συνέχεια και σχέση μας με τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία. Ποια είναι λοιπόν η θεώρηση της ε, κατάστασης αυτής και της ασφάλειας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα λέω αυτά. Έχουν οριστεί σε λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, την παγκόσμια ασφάλεια και είναι και στην καρδιά, όπως σας είπα, της ε, πολιτικής μας για την ανατολική ε, εταιρική σχέση και γειτονία. Πριν από ένα χρόνο η κυρία Μογκερίνη παρουσίασε τη συνολική αυτή στρατηγική. Σε αυτή τη νέα φάση της παγκόσμιας πολιτικής θα πρέπει η Ευρώπη να είναι στο ύψος των ευθυνών τη. Είναι ο βασικός, ο βασικός πάροχος ασφαλείας στην περιφέρεια. Είδαμε τα πρώτα φιλόδοξα αποτελέσματα μετά την παρουσίαση της στρατηγικής αυτής, μεταξύ αυτών μια μόνιμη στρατιωτική δομή για ε, την ε, διεξαγωγή μη εκτελεστικών ε, επιχειρήσεων και αποστολών. Τώρα θέλουμε από κοινού να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να έχουμε πιο αποτελεσματική δράση και στις αμυντικές δαπάνες με μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και ένα ταμείο αμυντικό που θα υποστηρίζει την έρευνα, την ανάπτυξη και την κοινή προμήθεια υλικού. Η Ένωση καλείται να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο και πιο ενεργό εκτός από την άμεση γειτονία της γενικότερα. Παράλληλα, η συνεργασία με το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι μεγάλη προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένα ε, αντιμετώπισε ένα αίτημα από όλους ενεχομένους να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στην ασφάλεια. Αυτό σημαίνει σταθεροποίηση ε, της περιοχής. Μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Και αυτή η αναθεωρημένη πολιτική έχει σημαντικό κεφάλαιο την ασφάλεια παραμένει ένας στόχος ανατολική γειτονία, όπω όπως ε, αναγνωρίστηκε σύνοδο κορυφή στη Ρήγα το 2015. Η διάσταση αυτή της ασφάλειας βασίζεται σε μια ει βάθος ανάλυση των παραγόντων ε, αποσταθεροποίηση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, σε κοινούς στόχους, κοινά συμπεφωνημένους στόχους, μαζί με τους εταίρους μας. θα πρέπει πάντα να συμβόμαστε στη συνεργασία τη θεμελιώδεις αρχές, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την χρηστή ε, διακυβέρνηση ε, και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχομαι λίγο τώρα στις σειράξεις που παραμένουν προφανώς το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία στο ε, μετασοβιετικό χώρο. Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες για να διαχειριστούμε και να επιλύουμε τις κρίσεις. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς ε, στηρίζουμε το διάλογο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις συγκρούσεις στην Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Ουκρανία, έτσι ώστε να βρεθούν ειρηνικές ε, και βιώσιμες λύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπροεδρεύει στη Γενέβη στην υπόθεση της Γεωργίας για να συνεληθεί ε, το θέμα ε, με ε, διαπροσωπικές επαφές σε όλη τη Γεωργία. Έχουμε στείλει και αποστολές στην Απχαζία και την Νότια Οσετία και παρακολουθούμε την κρίση στη Γεωργία και στον Κάφκασο σε συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερομένους. Αυτό είναι κάτι... Τώρα, Μολδαβία. Μετά από την μεταβατική περίοδο επίσης έχουμε υποβάλει προτάσεις οι οποίες στόχο έχουν να λύσουν τα επιμάχα Μετά από διάφορα μέτρα που θα χτίσουν εμπιστοσύνη, εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες της Γερμανικής και Αυστριακής Προεδρίας για τις ε, συνομιλίες. Τώρα, περνάμε στην, ε, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Εδώ υπάρχει μία έντονη κλιμάκωση το περασμένο έτος και εμείς συνεχίζουμε να καλούμε για κατάπαυση πυρός, να αρχίσουν ουσιαστικές συνομιλίες προς μια ειρηνευτική διαδικασία. Έγιναν πολλές και συχνές επισκέψεις ε, εκπροσώπων μας στην περιοχή που στηρίζουν τις προσπάθειες ε, των ε, συμπροέδρων. Περνάμε τώρα στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις μας όλο και εμβαθύνονται και γίνονται στενότερες τα τελευταία χρόνια παρά τις συνεχιζόμενες απειλέ στην ασφάλεια. Εδώ είδαμε δύο πολύ σημαντικά ορόσημα. Η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων που ετέθησε ισχύ στις 11 Ιουνίου και η Συμφωνία Σύνδεσης η οποία ετέθησε ισχύ μόλις την περασμένη Παρασκευή. Η Ουκρανία συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, βαθιές μεταρρυθμίσεις σε όλο το οικονομικό και πολιτικό σύστημα και έχει στήριξη άνευ για τις προσπάθειές της και πιστεύουμε πως αυτό βοηθά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας στις εξωτερικές απειλές ή προκλήσεις. Δυστυχώς, η κατάσταση της ασφάλειας στην Ανατολική Ουκρανία παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη και μία πλήρης ε, παρατηρητήριο για την κατάπαυση πυρός ε, δεν μπορεί να ε, γίνει μέχρι τώρα. Πέραν αυτού έχουν γίνει βήματα και από τις ε, δύο πλευρές τους τελευταίους μήνες για ε, να συνεχιστεί δυστυχώς η απομόνωση των κατοίκων της περιοχής αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να καλεί για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και θα συνεχίσει να στηρίζει την απόλυτη εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ και τις ε, προσπάθειες ε, σύμφωνα με το πρότυπο της Νορμανδίας. Και ε, επίσης θα συνεχίσει ότι η Ρωσία έχει υποχρεώσεις. Αυτό είναι κεντρικό στοιχείο της πολιτικής μας. Είμαστε όμω πρόθυμοι να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Όπω ανέφερε και είπατε εκπρόσωπο η κυρία Μογκερίνη, είμαστε πρόθυμοι να αυξήσουμε την υποστήριξή μα για την υλοποίηση και εφαρμογή των συμφωνιών ε, του Μίνσκ, αλλά και για την ανοικοδόμηση. Αυτή τη στιγμή στο επιτρέψουν οι συνθήκε. Βεβαίω θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε και να μην αναγνωρίζουμε την ε, ε προσάρτηση τη Κρυμαία και τη Σεβαστουπόλεω για την ε, Λευκορωσία. Την τελευταία δεκαετία οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας χαρακτηρίστηκαν από ένα κύκλο ελπίδας, απογοήτευσης και περιοριστικών μέτρων. Προσφέραμε τη συνεργασία μας ουσιαστικά μετά τα αποτελέσματα των εκλογών και επιβάλαμε περιοριστικά μέτρα όταν το Μίνσκ απέφυγε, ε, απέτυχε μάλλον να ε, ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις και προδιαγραφές. Ε, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε βελτίωση. Συμμετέχει περισσότερο στην ανατολική γειτονία η χώρα ή ακόμα έχουν αρχίσει και διαπραγματεύσεις για διευκόλυνση θεωρήσεις διαβατηρίων και πανεισδοχής. Επίσης ε, προχωράει μια ε, συμφωνία για ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στα ενεργειακά. Ένα σημαντικός νέος παράγων ήταν η περιφερειακή διάσταση που άλλαξε και ε, τη κατάσταση στην Ουκρανία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Λευκορωσία ήταν πολύ επικοδομητική σε αυτή την περίπτωση και επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει στην εσωτερική ακαιρεότητα ε, της Ουκρανίας και πάνω από 160.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν ε, εγκατασταθεί στη Λευκορωσία που τους υποδέχθηκε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τις σχέσεις μας ε, σε συνεργασία πάντα με μια επικριτική ματιά και σταδιακά βήμα-βήμα. Προχωρώ τώρα σε πιο συγκεκριμένα θέματα ασφάλειας, για το πώς ενισχύεται η ασφάλεια, η ε, αντοχή και το γεφύρωμα των ε, χασμάτων που υπάρχουν. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις κοινωνίες για να μπορούν να αντέχουν και να αντιστέκονται και στην Ανατολή και στο Νότο της Ευρώπης. Αυτή είναι μια στρατηγική που έχουν εγκρίνει και τα κράτη-μέλη ως βασική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης για να προχωρήσουμε σε μια προσέγγιση πιο διαφρομένη, πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του κινδύνου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ρόλο με τρεις τρόπους. Πρώτον, με διμερή συνεργασία, δεύτερον, διάλογο σε διμερή θέματα και τρίτον, να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο η εξωτερική πολιτική της Ένωσης μπορεί να συνεισφέρει στην αντοχή, στην αφεκτικότητα της ίδιας της Ένωσης, όχι μόνο των εταίρων. Ε, εδώ αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κοινό συμφέρον στο να απαντούμε συλλογικά ε, σε υβριδικές μορφές απειλής, κυβερνοτρομοκρατία, ε, και εξερμισμό και άλλα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, τις ρίζες του κακού και κάθε ε, πηγής ε, ανασφάλειας. Η πρώτη έκθεση για την εφαρμογή όλων αυτών δημοσιεύθηκε το περασμένο Μάιο και τονίζει τις κοινέ προσπάθειες που βάλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανατολική της εταίρη στην ασφάλεια. Αναγνωρίζει τις μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή η σύραξη στην Ουκρανία έχει επιδεινωθεί με μαζική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Εκτός από τις ή περίπλοκες λεγόμενες υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει χώρα. Τμήμα του ρόλου μας στην αντιμετώπιση όλων αυτών είναι η σωστή πληροφόρηση του κοινού. Γι' αυτό δημιουργήσαμε μια ε, για την Ανατολική Γειτονία, μια task force για να αποδομή, την ε, αποπληροφόρηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις χώρες ε, της Ανατολικής Γειτονίας. Θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει και τι ε, σημαίνει για τους πολίτες. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι διαπαιδαγώγηση των πολιτών για τα ευεργετήματα ε, και το όφελος που θα έχουν οι χώρες αυτές να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος δικαίου. Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δημιουργία θέσεων απασχόληση, ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς ε, θεώρηση διαβατηρίων. Αυτές ε, οι καμπάνιες σε όλες αυτές τις χώρες, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, ε, κλπ. έχουν ε, αυξήσει τη συνειδητοποίηση του κόσμου για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πολέμηση των απειλών στο διαδίκτυο, όπως είδαμε, αυξάνονται οι επιθέσεις και πολύ γρήγορα συνιστούν σημαντική απειλή για την ασφάλειά μας και την ευημερία μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεργάζεται με τις χώρες Ανατολικής Γειτονίας για να ενταθούν οι προσπάθειες και οι δυνατότητες της ε, ποινική δικαιοσύνης. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης χώρες αυτές, που σημαίνει και σταθεροποίηση των χωρών, αλλά και αξιόπιστους ε, θεσμούς. Έτσι οικοδομείται και εμπιστοσύνη με τα διάφορα μέτρα αυτά. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα διέπεται από την αντίστοιχη πολιτική μας. Ε, άλλο παράδειγμα, καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, της καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες και για την εσωτερική μας ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, για ε, την επιβολή του νόμου και τη σχετική κατάρτιση είναι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθούν στις χώρες αυτές για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης συνεισφέρει σημαντικά για την εφαρμογή ε, του ολοκληρωμένου τρόπου διαχείρισης και ελέγχου των σύνορων, ιδιαίτερα στα εξωτερικά ε, σύνορα με την Μολδαβία. Επίσης καταπολεμούμε το κυβερνοέγκλημα ιδιαίτερα στην Ουκρανία και έχουμε και επιχειρησιακή ετοιμότητα εκπαιδεύουμε διπλωμάτες, συνεργαζόμαστε στενά με τους ε, ε, ειδικού μας εντεταλμένους εκπροσώπους και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας δώσω για συγκεκριμένες δράσεις. CBRN, για τον περισμό του κινδύνου χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων, ε, καταπολέμηση ε, φυσικών καταστροφών και θεομηνών. Το 2017 έγινε και μια σχετική άσκηση. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω και την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, όπου συνεργαζόμαστε στρατηγικά και με το ΝΑΤΟ. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη Ρωσία και το ΖΑΠΑΤ. Η ενίσχυση λοιπόν της αντοχής αυτών των χωρών θα πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Επομένως, η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαία από πλευρά τη Ρωσίας, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η αποσταθεροποίηση της Ανατολική Ουκρανίας, εκτός από την υποδάβληση ε, παρατεταμένων σειράξεων γενικότερα στην περιοχή, είναι ε, επιβαρυντικοί παράγοντες. Υπάρχουν βασικά ε, σημεία, βασικές αρχές τελική πράξης του ε, Ελσίνκη που διέπουν τον ΟΑΣΕ. Ότι τα κράτη είναι κυρίαρχα, είναι ίσα και ε, διαμορφώνουν ανεξάρτητα όπως επιθυμούν τις σχέσει του με τις ε, άλλες ανεξάρτητες χώρες. Τα σύνορα είναι απαραβίαστα καθώς επίσης και η εδαφική ακαιρεότητα των κρατών. Είναι αναπόσπαστο δικαίωμα κάθε χώρας να αλλάζει τις συμφωνίες ε, ή την πολιτική ασφαλείας της. Εμείς θέλουμε να έχουμε συνεργασία με τη Ρωσία, επικοδομητική και παραγωγική, με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά βασική μας θέση είναι ότι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στη στάση μας απέναντι στη Ρωσία είναι να εφαρμοστούν πλήρως οι συμφωνίες του Μίνσκ. Αυτό ήταν και τμήμα της προσέγγισης που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το Μάρτιο του 2016, καθώς επίσης θέλουμε να βοηθήσουμε ε, τις χώρες αυτές να ενισχυθούν, να αυξήσουν την αντοχή τους, την αθεκτικότητά τους, άρα και τη δική μας. Σε ό,τι αφορά την άσκηση ΖΑΠΑΤ, πιστεύουμε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα ε, να κάνει ασκήσεις και με συμμάχους όταν αυτά γίνονται με τρόπο διαφανή σύμφωνα με διεθνείς κανόνες μεταξύ αυτών και των αρχών του ΟΑΣΕ που παραμένει η Ρωσία μέλος του. Τέλος για την Κεντρική Ασία. Είμαστε αναφαδόν υπέρ της περιφερειακής συνεργασίας που χρειάζεται οπωσδήποτε στην περιοχή για να αντιμετωπίσει και την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την συλλογική ε, περιφερειακή διαχείριση των φυσικών πόρων. Διασυνορική συνεργασία λοιπόν, εσωτερικές σχέσεις και θα πρέπει να επανασυνδεθεί το Αφγανιστάν με ε, μεταφορές, ενέργεια και εμπόριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να ενισχυθεί η ασφάλεια και τελικά η ευημερία στην περιοχή. Συμπέρασμα. να σα εξηγήσω πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα ασφάλειας στη μετασοβιετική εποχή, στο μετασοβιετικό χώρο. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στην Ανατολική ε, γειτονία και στην Νότια γειτονία. Υπάρχει χώρος για μεγαλύτερη συνεργασία και ανάγκη να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς εκεί. Με διεθνείς οργανισμούς και με τον ΝΑΤΟ. η χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα σύστημα με λογοδοσία έχουν καλύτερα αποτελέσματα και μπορούν να βοηθήσουν να προλαμβάνονται ένοπλες σειράξεις. Γι' αυτό έχουμε και την προσέγγιση αυτή απέναντι σε χώρες που θέλουν να μεταρρυθμιστούν με σωστούς θεσμούς, με χρηστή διακυβέρνηση και σεβόμενες τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι χώρες αυτές έχουν την υποστήριξή μας από την ίδια την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες στα κράτη-μέλη, ε, δεν ε, γνώρισαν ε, πόλεμες σειράξεις. Παραμένουν όμως οι σειράξεις είτε παγωμένες στην Ανατολή, είτε παρατηνόμενες, είτε θανατηφόρες. Άρα θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και πολυεπίπεδες δράσεις. αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας παράγον που εξασφαλίζει ακριβώς την ασφάλεια και την θα είμαστε στο σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεφίδα. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο James Σέρ για να μας παρουσιάσει τη δική του οπτική γωνία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ ενώπιόν σας, που με ξανακαλέσατε στην Επιτροπή σας δεύτερη φορά. Δύο μήνες μετά από τον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας, σε ένα γεύμα στην ε, Ρωσία, στη Μόσχα, ο πρόεδρος Μετβέντεφ είπε τα ακόλουθα. Αυτό είναι το δικό μας ε, κομμάτι, δική μας γωνιά του κόσμου. Με τους γείτονες μας συνδέει ιστορία, πολιτισμός και η ψυχοσύνθεση. Και επί 15 χρόνια σας λέμε πως δεν ανήκετε εδώ. Και σήμερα σας λέω πως δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτό. Και το επαναλαμβάνω, δεν θα το ανεχτούμε. Αυτό πριν το 1924. Πριν το 1924 η Ρωσία θεωρούσε πως ε, είχε στρατηγική αντεπίθεση εναντίον της 25χρονης γεωπολιτικής συμπεριφοράς φετερισμού της ε, Δύσης. Αυτά έχουν ακουστεί και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές συζητήσεις. Η Ρωσία όμως σε δημόσια λέει πως δεν έχουμε πρόβλημα με την Δύση όπως έχει παρουσιαστεί στην ιστορία. Αυτό που έχω, που, αυτό που είναι πρόβλημα όμως είναι πως ε, αμφισβητούν την πολιτική Δύση. Και αυτό έχει προεκτάσεις που φτάνουν μέχρι και τα σύνορα της Ρωσίας. Αυτό μάλιστα είναι αυτό που αποκαλούν οι Ρώσοι «Ρούσκι Μύρ», ο ρωσικός κόσμος. Κάτι το οποίο έχει τονίσει επανειλημμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ρωσικός κόσμος είναι πέρα από τα σύνορα ε, του ρωσικού κράτους ε, και είναι πέρα από το ρωσικό έθνος. Είναι ένας χώρος ο οποίος ιστορικά επηρεάζεται από τη Ρωσία. Από το 2008 η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατιωτική βία για να αλλάξει τα σύνορα. Και η κύρια διαμάχη που έχει είναι με τα πολιτικά σύνορα της Ευρώπης και όχι με τα φυσικά σύνορα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως πιστεύει πως η διάδοση της δημοκρατίας, της οικονομίας, της αγοράς, του κράτους δικαίου όπως ε, υπάρχει στην Ευρώπη είναι προς το συμφέρον όλων. Όμως η ρωσική ελίτ διαφωνεί και έχω μεγάλες αμφιβολίες ε, και δεν πιστεύω πως ε, θα αλλάξει κάτι με τον διάλογο. Θεωρώ επίσης απόλυτα σχετικό ότι αυτή η διάσταση του πολιτισμού ενισχύεται από τις γεωπολιτικές απόψεις του στρατιωτικού κατεστημένου της Ρωσίας. Διότι το στρατιωτικό αυτό κατεστημένο, κάτι που δεν είναι καινούριο, είναι πρακτική αιώνων, πριν ακόμα το 1917. Ορίζει την ε, απειλή διαφορετικά. Ορίζει την στρατιωτική πραγματική απειλή ως, ε, ε, ε, με βάση την εγκύτητα και τον χώρο και όχι με βάση την πρόθεση. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν σφαίρες επιρροής, υπάρχουν ενδιάμεσες ζώνες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ρωσική γεωπολιτική σκέψη. Και μάλιστα δεν έχουμε δει από τον καιρό του Μπρέσνιεφ και έπειτα μεγαλύτερη σύγκληση πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στο ρωσικό κράτος. Αυτή είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να παραδεχτούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει στην Ανατολική γειτονία. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, το πρόβλημα είναι ότι η Ανατολική γειτονία δεν είναι χώρος, αλλά είναι ένα σύνολο χωρών χώρες οι οποίες έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες και τα δικά τους συμφέροντα. Και πολλές από τις ε, χώρες αυτές θεωρούν ως ε, πρωταρχικό του στόχο τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Το πρόβλημα όμως είναι πως η Ρωσία θέλει να ορίζει εκείνη το τι σημαίνουν αυτές οι σχέσεις και η βασική έκφραση που χρησιμοποιεί η Ρωσία είναι με τους δικούς μας όρους. Η Αρμενία έχει αποφασίσει ότι το δικό της συμφέρον έχει ως εξής. Είναι πιο ισχυρή συμμετέχοντας σε διεθνείς συνθήκες, αλλά θεωρεί επίσης πως τα συμφέροντά της θα εξυπηρετηθούν καλύτερα από μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το φθινόπωρο του 2013 ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε σαφές με άκομψο τρόπο, το άκουσα και εγώ επανειλημμένα, Είπε λοιπόν στον πρόεδρο Σαρξιάν ότι αυτή η επιλογή δεν υφίσταται. Και τους έδειξε το πλωστάσιο που είναι διατεθειμένο να αγοράσει από τη Ρωσία το Αζερμπαϊτζάν και τους ρώτησε κατόπιν τούτου ποια είναι η δική σας απόφαση. Όταν ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς ήταν πρόεδρος της Ουκρανίας, αποφάσισε με δική του θέληση ότι στόχος της προεδρίας του είναι η Ουκρανία να μην ανήκει σε κάποιο μπλοκ και να παγώσει ως εκ τούτου τις ε, σχέσεις της με το ΝΑΤΟ έτσι ώστε να δεχτεί όλους τους όρους της ε, Ρωσίας για τον ε, ναυτικό στόλο στην Κρυμαία. Και κάνοντας αυτό θεωρούσε πως έτσι θα δημιουργήσει έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσε να καλλιεργήσει σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε λοιπόν να αυξάνεται η πίεση παντού μέχρι και στη δημόσια τηλεόραση όταν ο Βίκτορ Γιαννουκόβιτς είπε ε, ότι ζητάτε πολλά και ο, η απάντηση που έλαβε είναι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Και λίγο πριν την απόφαση του να σταματήσει τις ε, διαπραγματεύσεις, να σπάσει τη συμφωνία σύνδεσης, ο πρόεδρος Πούτιν του υπαγόρευσε με κάθε λεπτομέρεια το πόσο εύκολο είναι η Ρωσία να διαλύσει την οικονομία της Ουκρανίας και να κρατήσει τον ε, πρόεδρο Γιανουκόβιτς υπόλογο γι' αυτό. Τώρα, εάν αυτό ήταν μπλόφα ή όχι, είναι άλλη ερώτηση, αλλά τα γεγονότα ήταν αυτά. Τη δεκαετία του 90 είχα στενή συνεργασία με την ε, διπλωματία και του ε, υπεύθυνου για την άμυνα της Ουκρανίας και βλέπω πω σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα αυτό που τότε συζητούσαν θεωρητικά. Ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα η Ουκρανία μετά από καθημερινή πίεση από τη Ρωσία αναγκάστηκε να κάνει βήματα ενάντια στο δικό της συμφέρον. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο των ε, ρωσοουκρανικών σχέσεων. Γι' αυτό λοιπόν δεν ε, είναι δικές μου εικασίες αυτά. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν από τη δεκαετία του 90. Και θα έλεγα συμπεραίνοντας πως ε, παρότι δεν βλέπω σήμερα κάποια ένδειξη για το ότι η Ρωσία επανεξετάζει τα συμφέροντά της στην περιοχή αυτού που ονομάζουμε εμείς Ανατολική Γειτονία, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όπως αναθεωρεί μεν τη στρατηγική της, δεν γνωρίζει δε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά της. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Υπάρχει ένα αδιέξοδο στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, όχι εξαιτία της δυτικής πολιτικής, αλλά εξαιτία της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας, η οποία απεδείχθη πολύ δυνατότερη από αυτό που περίμεναν. Και παρότι δεν μου αρέσει ούτε εμένα να το λέω ούτε και σε εσά να το ακούτε, ο κύριος λόγος της προσοχής της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση Τραμπ. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτό που λέμε ζαπουτσιόνικα, φυλακισμένος, κρατούμενος. Ανάμεσα στην κυβέρνησή του, στην αμυντική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών και ανάμεσα σε εκείνου ε, που αποτελούν τους συνεργάτες του. Και μάλιστα το επιτελείο του Τραμπ είναι πολύ σκληρότερο στη στάση του απέναντι στη Ρωσία από ότι το επιτελείο του Ομπάμα. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έχει δείξει πως είναι έτοιμοι για δράση όταν καταπατώνται κόκκινες γραμμές, πως είναι σε θέση μονομερός, χωρίς προειδοποίηση, να δράσει. Και παρά το γεγονός ότι αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για την Ευρώπη, η αλήθεια είναι πως ε, είναι κάτι που περιορίζει τη Ρωσία. Και υπάρχουν μάλιστα και παραδείγματα στη Συρία για τη στάση αυτή. Έχουν γίνει προσπάθειες λοιπόν να αλλάξει η Ευρώπη εκ των έσω, έχουν γίνει προσπάθειες παρέμβασης στα εκλογικά ε, συστήματα και στις εκλογές σε χώρες της Ευρώπης, τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν τα επιθυμητά. Και τέλος, θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι... Εμείς, προσπαθούμε σε αυτή τη γωνιά του κόσμου να καταλάβουμε τι συμβαίνει από την δική μας οπτική γωνία, από την ε, οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σοβαρή γεωπολιτική δύναμη. Και είναι καιρός να το αναγνωρίσουμε. Το δεύτερο συμπέρασμα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω προς ε, προβληματισμό είναι ότι οι αντιλήψεις αυτές είναι βαθιά ριζωμένες στο ρωσικό λαό. Δεν είναι η άποψη του Βλαντιμίρ Πούτιν μόνο. Και ακόμα και κάτω από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες, και να πω εδώ ότι οι συνθήκες είναι δυσμενείς, μετά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και γνωρίζω πως στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Ρωσία είχε πολύ διαφορετική προοπτική. αν μάλιστα μία ρομαντική αν θέλετε περίοδο. Αυτό όμως άλλαξε πολύ νωρίς και μάλιστα πολύ πριν το συνειδητοποιήσουμε εμείς. Τέλος. Να πω ότι Ω εκ τούτου, η ανατολική γειτονία και η σχέση μας με αυτή θα πρέπει να επιβιώσει συνθήκων άκρο ανταγωνιστικών. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, τι θα έπρεπε να κάνουμε και τι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να κάνουμε. Και μια και μου μένουν 45 δευτερόλεπτα να δώσω και ένα τελευταίο ιστερόγραφο αν θέλετε για το ΖΑΠΑ 2017. Ίσως, εάν επαληθευτούν οι υποψίες μου, θα είναι μια μεγάλη ενέργεια αποκλιμάκωσης. Εάν αναλογιστούμε τις χειρότερες συνέπειες, δεν θα μας βοηθήσει. Δεν θα μας βοηθήσει εάν η προσοχή αλλάξει και δοθεί έμφαση σε αυτά που μόλις σας είπα. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. <laughs> And now I kindly ask Professor uh, Andres to take Ο κύριος Ράτς έχει το λόγο, καθηγητής Ράτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι για δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω ότι αυτά τα οποία θα σας πω είναι αυστηρά προσωπικές μου απόψεις. Δεν εκπροσωπώ κανένα κράτος ή διεθνή οργανισμό ή οποιαδήποτε μορφη οργάνωση. Είναι και βολικό και άβολο να μιλάει κανείς μετά από τον James Σαρ. Θα μπορούσα να σταματήσω να μιλάω από εδώ και πέρα. Όμως θα προσθέσω κάποιες λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ κυρίως στα θέματα της Ουκρανίας, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Γιατί η Ρωσία θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι από πλευράς ρωσικής προοπτικής η χρήση των ενόπλων δυνάμεων και όπλων για πολιτικούς στόχους είναι μια success story από το 2008. Το έκαναν στην Γεωργία και αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα μπορέσει τελικά από ό,τι φαίνεται να μπει στο ΝΑΤΟ η Γεωργία. Στην Ουκρανία από το 2014 και μετά πέτυχαν ακριβώς τους ίδιους στόχους σε σχέση με την Ουκρανία και εξασθένησαν θα έλεγα και ε, αποδυνάμωσαν την Ουκρανία για δεκαετίες ολόκληρες. Ε, ξεκίνησαν και την ένοπλη παρέμβασή τους το 2015 στην Συρία. Να πω εδώ ότι είναι η πρώτη διεθνής παρέμβαση, μίζων διεθνής παρέμβαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Η επιχείρηση στη Συρία κατάφερε να καταστήσει την Ρωσία μια ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη και αύξησε το ρόλο της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την έβρεση λύση στο Συριακό. Γι' αυτό λοιπόν μετά από όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα σταματήσει η Ρωσία αυτή την πρακτική. Θα χρησιμοποιεί πάντα στρατιωτικές δυνάμεις για πολιτικούς στόχους. Το θέμα δεν είναι, πολιτικέ, είναι στρατιωτικές συγκρούσεις ή στρατιωτική επικράτηση, το θέμα είναι πολιτική διελκυστίνδα. Δεύτερον, για το Ζαπάντα. Οι ε, ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι έτοιμες για μια παγκόσμια σύραξη. Να πω ότι η αρχική προθεσμία για τη μεταρρύθμιση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για το 2020 σε τρία χρόνια από τώρα δεν θα επιτευχθεί. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά εμπόδια στον δρόμο αυτό για τη μεταρρύθμιση των στρατιωτικών δυνάμεων. Υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης λόγω της ενδογενούς αδυναμίας της ρωσικής οικονομίας, της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Ε, να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάνω από 600 προγράμματα ε, στρατιωτικά στην Ρωσία που δεν μπορεί να ολοκληρωθούν γιατί εξαρτώνται από τη δυτική τεχνολογία σε μια δημοσίευση ενός ερευνητικού ιδρύματος στη Μεγάλη Βρετανία ε, τίθεται θέμα και για την ανεξαρτησία ε, και από την εξάρτηση των Ρώσων από την αεροπορική βιομηχανία της Ουκρανίας και για τα ελικόπτερα και τα μεταφορικά αεροσκάφη ε, και κινητήρες πυράβλων και άλλες μορφές κινητήρων. Υπάρχουν επίσης και οι γνωστές ε, ε, δημογραφικές ανησυχίες που υπονομεύουν την Ρωσία. Υπάρχει αυξημένη διαφυγή εσόδων λόγω λαθρεμπορίου, ναρκωτικών ή μη κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο ρωσικός στρατός κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να τις φέρει πέρας και αυτό το απέδειξε στη Συρία. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω ότι ο ρωσικός στρατός δεν είναι έτοιμος για μια παγκόσμια σύγκρουση. Να θυμηθούμε τους πολέμους τους οποίους διεξήγαγαν από το 2008 Γεωργία, Ουκρανία και Συρία. Οι πόλεμοι αυτοί διεξήχθηκαν εναντίον εχθρών ασθενεστέρων της Ρωσίας. Ε, συνεπώς λοιπόν μιλάμε για διαφορετική κλίμακα το να πολεμήσουν εναντίον του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στον Giles του Chatham House που είπε ότι οι δυνατότητες κινητοποίησης της Ρωσίας δεν συνοδεύονται, σε επίπεδο δηλαδή στρατιωτικού προσωπικού, δεν συνοδεύονται από τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Ένα πράγμα είναι να κινητοποιήσεις εκατοντάδες χιλιάδες στρατού και ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιήσεις όλες τις επιχειρησιακές σου ικανότητες. Σε έξι μήνες ε, στη Ρωσία επίσης έχουμε προεδρικές εκλογές. Δεν είναι η στιγμή κάποιος από τους εκπροσώπους της ελίτ της Ρωσίας να επιθυμεί ένα τέτοιο είδους πόλεμο. Σχετικά με την Ουκρανία τώρα. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω σαν πανεπιστημιακός ότι εμένω στα θέματα της ορολογίας και μιλάμε για την Ουκρανική σύραξη ή τη σύραξη στην Ουκρανία. Είναι δύο εκφράσεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Εγώ προτιμώ να μιλάω για την σύγκρουση στην Ουκρανία, τη σύραξη στην Ουκρανία. Όταν μιλάμε Ουκρανική σύγκρουση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι μια εμφύλια διαμάχη, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο πραγματικά. Είναι λοιπόν σωστό να μιλάμε για την σύραξη στην Ουκρανία. Είναι δύσκολο να κατηγοριοποιήσει κανείς τη σύραξη αυτή. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την ορολογία του Φρίντμαν που ε, θεωρεί ότι είναι ένας λεγόμενος περιορισμένος πόλεμος. Περιορισμένο σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές στην πρώτη γραμμή υπάρχει ένας ξεκάθαρος ανοιχτός πλήρης πόλεμος. Ταυτόχρονα όμως διεξάγονται διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες, είναι ανοιχτά τα σύνορα, υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές, υπάρχει λοιπόν ένας πόλεμος όχι για όλους, περιορισμένος λοιπόν, και τώρα είναι τρίτος χρόνος που διεξάγεται ο πόλεμος αυτός. Τώρα για τις ζώνες των συγκρούσεων. Να ξεκινήσω με την Κρυμαία για να είμαι σύντομος και κατανοητός. Μετά από την παράνομη κατοχή της Χερσονήσου, η Ρωσία έχει προχωρήσει στην έντονη στρατιωτικοποίηση της Κρυμαίας. Αυτό δεν έγινε για να αποκριστούν οι ουκρανικές επιθέσεις. Ανέπτυξε αμυντικές δυνάμεις ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης των αεροπορικών επιθέσεων και των ναυτικών επιθέσεων ενίσχυσε λοιπόν τις δυνατότητες της Χευσονήσου από πιθανές επιθέσεις από την Δύση. Τώρα είναι πολύ πιο ισχυρή η περιοχή ε, πολύ πιο ισχυρή από ότι αν φοβόντουσαν μόνο την ε, Ουκρανία. Η στρατιωτικοποίηση της Κρυμαίας συνοδεύεται δυστυχώς από μαζικές και συστηματικές παραβιάσεις ε, του πληθυσμού του τοπικού και των Ουκρανών και των Τατάρων. Ε, τα άσχημα νέα εδώ είναι ότι εφόσον η Ρωσία όπως γνωρίζουμε βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι προφανές ότι η κατάσταση στην Κρυμαία δεν αλλάζει. Σχετικά τώρα με την Ανατολική Ουκρανία ε, έχουμε να κάνουμε με μια ανοιχτή ε, σύγκρουση, δεν είναι παγωμένη όπως είχε υποθεί η σύγκρουση, παραβιάζονται οι ε, συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, υπάρχουν θύματα και από τις δύο πλευρές, δεν έχει καμία σχέση με την υπερνηστερία, πρόκειται για έναν περιορισμένο πόλεμο εν εξελίξη. Η ρωσική στρατηγική για την Ανατολική Ουκρανία έχει αλλάξει τέσσερις τουλάχιστον φορές πριν από την, από την αρχή του πολέμου. Στην παρούσα στιγμή φαίνεται ότι η Ρωσία προσπαθεί να διατηρήσει την περιοχή του Ντόνμπας μέσα στην Ουκρανία. Ε, κρατάει λοιπόν τις περιοχές αυτές ε, εντός της Ουκρανίας αλλά υπό ρωσικό έλεγχο και έτσι καθιστά την Ουκρανία ασθενέστερη και δυσλειτουργική σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τώρα συνέπειες. Οι ένοπλες δυνάμεις της λεγόμενης ε, δημοκρατίας του Ντονιέτσκα και της δημοκρατίας του Λουχάνσκα που δεν αναγνωρίζονται από κανένα, οι στρατιωτικές δυνάμεις αυτών των δύο οντοτήτων αντιπροσωπεύουν περίπου 40.000 ε, ε, στρατιώτες, 400 ε, τεθωρακισμένα, επίσης και αντίστοιχο αριθμό τεθωρακισμένων μεταφοράς και επίσης εκπαίδευση των αξιωματικών των στρατών αρχών και όλα αυτά καθιστούν τις στρατιωτικές αυτές δυνάμεις διαλειτουργικές με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Είναι δηλαδή ρωσικές δυνάμεις δι' αντιπροσώπου ουσιαστικά. Ο στρατηγικός στόχος της ρωσικής πλευράς είναι στην ουσία να διαβεβαιώσουν ότι η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να τερματίσει τη σύγκρουση στρατιωτικά από μόνη της. Ακόμα και αν η Ουκρανία πάρει ας πούμε αντιαρματικά όπλα από τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα αλλάξει η ισορροπία των δυνάμεων. Αυτά ήταν τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σήμερα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές τις οποίες είχε στη διάθεσή της η χώρα του 14. Σαν πανεπιστημιακόν μου αρέσει να διαβάζω. Και γι' αυτό θα διαβάσω από ένα πολωνικό βιβλίο εξαιρετικό του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών και λέγεται το άρθρο ο, στρα... ο ισχυρότερος στρατός τον οποίο έχει ποτέ η Ουκρανία. 200.000 προσωπικό και με πάρα πολύ μεγάλη στρατιωτική εμπειρία. <clears throat> Έκανε κάτι το χωρίς προηγούμενο. Όλες οι μονάδες μάχης πέρασαν από την πρώτη γραμμή, ενάλλαξαν η μία την άλλη και απέκτησαν έτσι α, εμπειρία στον τομέα της μάχης. Σκεφτείτε πόσες από τις δικές σας μονάδες, τους δικούς σας στρατούς έχουν εμπειρία πολεμική. Η Ουκρανία όλοι. Είναι σε θέση λοιπόν να διατηρηθούν στην πρώτη γραμμή <clears throat> εναντίον των ε, ρωσικών δυνάμεων και των ε, ακολούθων ε, των Ρώσων, αυτών που θέλουν να αποσχιστούν και αυτό έχει αλλάξει από το 2014 μέχρι τώρα. Οι επιθέσεις που έγιναν λοιπόν το τελευταίο καιρό ε, θα έλεγα αντιμετωπίζονται από τον Ουκρανικό στρατό, υπάρχει μια σταθερότητα, το ηθικό είναι ιδιαίτερα υψηλό του Ουκρανικού στρατού και αποκτάται συνεχώς ε, εμπειρία πολεμική. Είναι σε θέση να διεξάγει επίσης και αποστολές μυστικές πέραν της γραμμής των αποσχιστικών ρωσικών δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ξεκάθαρη βέβαια πολεμική, πλήρης πολεμική σύραξη ανοιχτή από πλευράς ιδιαίτερα Ρωσίας. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται βέβαια στην περιοχή επηρεάζουν και την ίδια την Ουκρανία. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι οι στρατιώτες και οι κρατούμενοι που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες που υποφέρουν από μετατραυματικά ψυχολογικά θέματα και δεν έχουν ιδιαίτερη βοήθεια. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το μέλλον. Η διαφθορά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική στην περιοχή και συνεχίζεται. Για να σας δώσω κάποια επίσημα στοιχεία που τρομάζουν, το 2016 οι απώλειες των μαχητών, των μη μαχητών μάλλον, του Ουκρανικού στρατού είναι υψηλότερες από τους μαχητές. Δηλαδή, ε, αυτοκτονία, δολοφονίες, ατυχήματα οδικά, μεθυσμένοι. Ε, δηλαδή, τα θύματα από τέτοιες δραστηριότητες είναι πιο πολλά από τα θύματα στην πρώτη γραμμή, από την πολεμική σύραξη αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως ότι η Ρωσία, επαναλαμβάνω, είναι σε θέση, ή είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει εναντίον της Ουκρανίας έναν ανοιχτό πλήρη πόλεμο. Και νομίζω ότι θα μπορούσε και σε ένα μεγάλο βαθμό, αν κάτι τέτοιο δυστυχώς συμβεί, να αντισταθεί. Τώρα, αν δώσουμε ισχυρά όπλα, αυτό θα αυξήσει το τίμημα για το Κρεμλίνο, ακόμα και αν αποφασίσει μια τέτοια μαζική επίθεση και νομίζω ότι αυτό σκέπτονται και οι Αμερικανοί ότι ενισχύοντας αποτρέπουν. Τώρα από το 2018 υπάρχουν και κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία και είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμα και αν ε, βρισκόμαστε λίγο πριν από τις ρωσικές προεδρικές εκλογές, δεν περιμένω την Ρωσία να κάνει σύντομα κάτι το σημαντικό στην Ουκρανία διαφορετικό από αυτά τα οποία κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα, η κατάσταση στις διμερείς σχέσεις ε, μπορεί να γίνει, θα έλεγα, πολύ πιο ευαίσθητη και σας ευχαριστώ. I ask, ε, Ευχαριστώ. Τώρα θα πάρει το λόγο η κυρία Μαρία Δίνερ για να μας παρουσιάσει το θέμα της. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, ε, που είναι η δεύτερη που μου απευθύνεται. Επειδή και οι προλαλήσανες μίλησαν και οι δύο αγγλικά, θα μιλήσω και εγώ αγγλικά. Στην αρχή ήθελα να μιλήσω πολωνικά, αλλά δεν ξέρω πώς είναι καλύτερο για όλους να μιλήσω αγγλικά. Present, um... Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για τις εξελίξεις στην ασφάλεια στη Λευκορωσία, μεταξύ αυτών και ε, στη, ε, στις ένοπλες δυνάμεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις ε, ΖΑΠΑΤ, Δύση. ήθελα αρχικά να σας πω το εξής προσάρτηση της Κρυμαίας και ο πόλεμος στην Ανατολική Ουκρανία τι έδειξαν. Ότι η στρατηγική, η αρχιτεκτονική καλύτερα ασφαλείας στην ε, Ανατολική Ευρώπη έχει πρόβλημα. στο παρελθόν ασχολούμασταν στη Ρωσία με τις μυστικές υπηρεσίες, την ΚΑΓΕΜΠΕ και άλλα και τώρα με τις ένοπλες δυνάμεις. Έχει αλλάξει η Λευκορωσία έχει αλλάξει και στρατιωτικό δόγμα το από τον Ιούλιο 2016 ε, μετά από την αλλαγή της πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης στην Ανατολική Ευρώπη. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι αυτό το στρατιωτικό δόγμα που εστιάζει και στις υβριδικές απειλές αλλά και στον ε, ηλεκτρονικό πόλεμο των πληροφοριών. Και οι απειλές αυτές δεν είναι απειλές ε, ε, εκδισμών, αλλά εξανατολών. Ενδιαφέρον στοιχείο. Τι γίνεται τώρα με τις ένοπλες δυνάμεις στη χώρα, ελπίζω να βλέπετε τη διαφάνεια πάνω κάτω. Τα τελευταία 25 χρόνια το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μειώθηκε τέσσερις φορές, στο ένα τέταρτο. 46.000 ε, έστολοι και 13.000 πολίτες υπηρετούν σε 8 ε, ε, σώματα που υπάγονται στο Υπουργείο Αμήνης της Δημοκρατίας Λευκορωσίας. Το 60% είναι επαγγελματίες με συμβάσεις και 40% είναι κληρωτοί είναι ε, η στρατιωτική θητεία υποχρεωτική, τουλάχιστον για 12 μήνες, ε, για πτυχιούχους και 18 μήνες ε, για μη πτυχιούχους. Βλέπετε εδώ πώς διαρθρώνεται ο στρατός δυτικά και βόρειο-δυτικά. Δεν υπάρχει σώμα στρατού προς Ανατολά, μόνο προ τη Δύση και το, το Βορρά. Καταλαβαίνετε η χώρα πώς προσανατολίζεται και πού είναι το ε, δόγμα της το στρατιωτικό στραμμένο. Συνεχίζω. Εδώ βλέπουμε τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. 515 άρματα μάχης, 827 ε, μονάδες πεζικού 240 ε, συστήματα εκτόξευσης πυράβλων ε, περιορισμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα αξιόμαχα, πράγμα που είναι προβληματικό γιατί εξαρτώνται απολύτως από τη Ρωσία και για την ε, άμυνά τους. Εδώ σε αυτή τη γραφική παράσταση βλέπετε ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι 1 με 1,5% μόλις. 500 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Που ήταν 4 με 5% του προπολογισμού. προφανές ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τη Ρωσία και με τον ΝΑΤΟ. Ούτε μπορούν να είναι ταυτόχρονα και με τον ΝΑΤΟ και με τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία με τη Ρωσία. Είναι ο βασικός πολιτικός, οικονομικός αλλά και ε, αμυντικός εταίρος και έχουν πολλών ειδών συμμαχίες με τη Ρωσία. Έχουν και οικονομική συμμαχία. Ε, και αν και θεωρητικά η Λευκορωσία είναι ε, ουδέτερη στρατιωτικά, συμμετέχει στην οργάνωση συλλογική συμμαχίας. Και τα δύο κράτη κάθε χρόνο έχουν κοινέ στρατιωτικές ασχήσεις που είναι γνωστές με τον όρο Ζάπα φετινή, ονομάζεται Δύση. Η περσινή έγινε ε, Μάλλον η τελευταία που έγινε ήταν το 2013, αλλά υπάρχουν και μεγάλες ε, ασκήσεις με το όνομα ε, Σπίδα της Ένωσης. Τελευταία άσκηση Ζάπατα έγινε το 2013, όπως σας είπα, στη Δυτική Λευκορωσία και στην επαρχία ε, του Καλίνιγκρατ. Και το σενάριο αντιμετωπίζει μάχες τύπου Αραβικής Άνοιξης. Οι αρχές της χώρας λοιπόν προσπάθησαν ε, και να αντιμετωπίσουν μια υποτιθέμενη ε, επίθεση ε, τρομοκρατών με 70 άρματα, με 60 ελικόπτερα και αεροσκάφη, με ε, συστοιχίες ε, πυράβλων και τα λοιπά. Και με ε, ταυτόχρονες ασκήσεις στη στόλου της Βαλτικής θάλασσας, του Ρωσικού. Αντίστοιχα και με την άλλη άσκηση Union Shield του 2015, πάλι το Σεπτέμβριο, 6.700 συμμετείχαν από τη Ρωσία και 1.300 στρατιωτικοί από την Λευκορωσία και με βαρύ οπλισμό, περίπου 400 όπλα. Συμμετέχουν στο πλαίσιο του ΣΥΣΤΙΟ και κάθε χρόνο διοργανώνουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Σερβία στην σλαβική ε, αδελφότητα όπως την ονομάζουν. Τι γίνεται με τη στρατιωτική εξάρτηση. Η Ρωσία εξαρτάται και αυτή σε κάτι από τη Λευκό-Ρωσία. από τη Σοβιετική εποχή αυτό χρονολογείται. Ε, στην παραγωγή ε, κάποιων πλατφορμών ε, για πυρηνικούς πυράβλους και μη πυρηνικούς που παράγονται στο Μίνσκ. Και κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Η Λευκορωσία μπορεί να εξυγχρονίζει κάποιους κινητήρες ε, σοβιετικούς, ε, ρωσικούς, ε, πράγμα που έκαναν μέχρι τώρα οι Ουκρανοί και για τα αεροσκάφη και για τα άρματα μάχης. Αλλά λόγω τώρα του πολέμου στην Ουκρανία αυτό έχει σταματήσει. Αν κοιτάξουμε στο χάρτη θα καταλάβουμε τι σημασία έχει η Ρωσία για τη Λευκορωσία και πόσο απέχει η Μόσχα από τα σύνορα του ΝΑΤΟ. Ε, και αυτό καθιστά τη Λευκορωσία πάρα πολύ σημαντική χώρα για τη Ρωσία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, από τη σκοπιά της Ρωσίας η Λευκορωσία είναι δικό τους έδαφος. Αυτό αφορά και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθετικές και τις αμυντικές. Και τολμώ να πω ότι από τη ρωσική σκοπιά η Λευκορωσία είναι Ρωσία, όχι η Λευκορωσία. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες για τα γυμνάσια Ζάπατ, Βλέπουμε τι έχει στις δυτικές περιοχές η Ρωσία. Δεν αφορά μόνο τους πυράβλους Ισκαντέρ, αλλά και κάποια υβριδικά συστήματα που έχουν ε, δοκιμάσει κατά τον πόλεμο στη Συρία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ε, υποβρύχια στη Βαλτική. Έχουν ένα βεληνικές 200 χιλιόμετρων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε τακτικές εχθροπραξίες και σε, και, σε τακτικά όπλα και σε πυρηνικά. Βλέπετε εδώ το χάρτη για το πώς ε, αλλάζει η κατάσταση στο ε, ανατολικό σκέλος. Η Ρωσία έχει αποφασίσει να μεταφέρει τρεις μεραρχίες ε, πράγμα που αλλάζει ε, τελείως την κατάσταση στα σύνορα. Άλλαξαν και το δόγμα λοιπόν προς τις μας και επίσης άλλαξε και η διοίκηση εντελώς του στόλου της Βαλτικής θάλασσας. Φέτος λοιπόν η ασκήση ΣΑΠΑΤ θα είναι και μια δοκιμή για τις ε, ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας για τη νέα στρατιωτική δομή για την πρώτη στρατιά και ε, θα δοκιμαστεί και η νέα διοίκηση του στόλου της Βαλτικής. Όπως γνωρίζετε, στην Λευκορωσία και τη Δυτική Ρωσία γίνονται οι στρατιωτικές αυτές ασκήσεις. Επίσημα ε, συμμετέχουν 20.700 στρατιωτικοί 13.000 Μάλλον είναι 12.700, 3.000 Ρώσοι και πρέπει να προσκαλέσουν υποχρεωτικά και παρατηρητές από τις χώρες του ΟΑΣΕ. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση αυτή. Οι ε, ασκήσεις αυτές είναι ένα τμήμα της ευρύτερης εικόνας και ε, θα κάνει ταυτόχρονα γυμνάσια και ο στόλος της Βαλτικής θάλασσας όπου θα δούνε και το αξιόμαχο και την υπηρεσιακή ετοιμότητά τους και στο, στη Δύση και στο Νότο. Δηλαδή η Ρωσία δεν προετοιμάζεται απλώς για να δραστοποιηθεί στη Λευκορωσία αλλά γενικότερα. Επίσης δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις ασκήσεις που γίνονται στη Δύση, Ζάπαν, αλλά και στο Ανατολικό ε, άκρο, γιατί είχαμε και κοινέ ασκήσεις πρόσφατα με τη Μογγολία. Τι, ποιες είναι οι προθέσεις της Ρωσίας να διατηρήσει κάποιες χώρες υπό τον έλεγχό της να αυξήσει την πίεση προς την Πολωνία και χώρες της Βαλτικής και το σενάριο που παρουσιάστηκε στο λαό την περασμένη εβδομάδα ήταν όταν, ότι η Λευκορωσία χρειάζεται τη Ρωσία για την άμυνά της και κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει η Λευκορωσία θέλει να προβάλλεται ως πιο ε, ειλικρινής και πιο διαφανής από τη Ρωσία αλλά Πώς εμείς θα τους θεωρήσουμε τέρο, αν εκείνοι μας θεωρούν το βασικό τους εχθρό. Αν κοιτάξετε το χάρτη των ασκήσεων, ε, οι δύο χώρες ε, προς οποίες, κατά τον οποίων στρέφεται είναι Πολωνία και Λιθουανία. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ποιες είναι οι προθέσεις τους και τι αποσκοπούν και σε τι αποσκοπούν μάλλον και γιατί θέλουν να συνεργαστούν. Συμπέρασμα. Η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι ρευστή ξέρουν ότι θα πρέπει να έχουν στη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον εταίρους, γιατί βγάλαν τα συμπεράσματά τους και τα διδάγματα από την κατάσταση στην Ουκρανία. Ε, διακατέχονται από μεγάλο φόβο μήπως απομονωθούν μόνο με την ε, Ρωσία, αλλά δεν θα πρέπει να περάσουν και τις κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές όμως και από την ε, Ρωσία και ε, από την συμμαχία και την οικονομική και τη στρατηγική με τη Ρωσία. Και προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Ρωσία ε, θα αφήσει στρατεύματα μετά τις ασκήσεις στην επικράτεια της Λευκορωσίας. Δεν χρειάζεται αυτό. Βλέπετε πώς έχουν αναθεωρήσει ε, ότι έχουν κοντά στα σύνορα μεραρχία τεθροκισμένων, έχουν κοινά συστήματα αμυντικά. Ε, ο στρατός Λευκορωσίας είναι πιο πιστός στη Μόσχα και λιγότερο στο Μίνσκ. Γιατί οι ψηλόβαθμοι αξιωματικοί, ανώτατοι αξιωματικοί ε, έχουν εκπαιδευτεί στην Μόσχα. Και όποιο έχει υπηρετήσει το στρατό τη Λευκορωσία μπορεί χωρί κανένα πρόβλημα να τα καταταγεί ή να ε, βρει απασχόληση με συμβόλαιο στο ρωσικό στρατό. Άρα υπάρχει ρωσικό έλεγχο εκεί πλήρη των ενοπλών δυνάμεων τη Λευκορωσία. Όπω είπε και ο άντρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Συνεχίζεται η μεταρρύθμιση και στο ρωσικό στρατό Ε, θέλουν ε, να εξακολουθούν να ελέγχουν τις χώρες που θεωρούν ότι είναι χώρος επιρροής τους. Ε, είναι σαφές αυτό και ακόμα και αν προσπαθήσουν οι Λευκορώσοι να έχουν μια συμπεριφορά του κράτους, είναι πάρα πολύ περιορισμένο το περιθώριο ελιγμών τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντίνε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο επικεφαλής διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Και θα ήθελα να τους δώσω το λόγο. Πρώτα στον κύριο Σδρογεύσκη, επικεφαλής της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας καταρχάς όλους. Άκουσα πολλά ενδιαφέροντα από τους ε, συμμετέχοντες, από τους προσκεκλημένους, ε, μια διάγνωση για την κατάσταση στην Ουκρανία, μια διάγνωση για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούστηκαν. Και πολύ ενδιαφέροντα ήταν επίσης και τα συμπεράσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Έχω την εντύπωση πως ε, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές τις περιοχές μαζί, συνολικά. Και επίσης να τις εξετάσουμε μαζί και την περίπτωση της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας και της ε, Γεωργίας γιατί νομίζω πως ε, συνδέονται άμεσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πάρα πολύ όλους. Νομίζω πως οι παρουσιάσεις ήταν πολύ καλές, αλληλοσυμπληρώθηκαν και έκαναν μια πολύ σωστή διάγνωση της κατάστασης. Αυτό όμως που παρατηρώ και με ανησυχεί είναι πως ελείπουν ακριβέστερες προβλέψεις για την κατάσταση στις περιοχές αυτές σε αυτήν εδώ την Επιτροπή πολύ συχνά ασχολούμαστε με το στοιχείο της έκπληξης και βλέπω πως υπάρχουν πολλές πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουμε από διάφορες πηγές και δεν έχουμε συνδέσει ακόμα. Εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι γίνεται με τις προβλέψεις σας. Υπάρχει κάποια πρόγνωση, μπορούμε να πούμε κάτι για το μέλλον, για το τι θα γίνει και στον στρατιωτικό τομέα και στην οικονομία και στην πολιτική αλλά και τον κυβερνοχώρο. Τι γίνεται με τις εχθρικές, με τις προπαγανδιστικές δραστηριότητες που ε, λαμβάνουν χώρα εκεί. Όπως ακούσαμε χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για προπαγάνδα και κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εμείς στην Ευρώπη ως απλοί παρατηρητές που δεν έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες, να περιμένουμε μέχρι να μάθουμε περισσότερα για το τι συμβαίνει ή μήπως οι δομές που έχουμε, τα προγράμματα, η συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είναι πιο επιθετικά, να προσαρμοστούν δηλαδή στη στάση της Ρωσίας. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο. Επικεφαλής της ε, Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την καταπληκτική επιλογή των ε, εμπειρογνωμόνων, πολύ ενδιαφέρουσες, εμπεριστατωμένες ε, ε, εισηγήσει, αναλυτικές, ε, μεταξύ τους αλληλοσυμπληρούμενες και ταυτόχρονα ανησυχητικέ. Ουσιαστικά, με άλλα λόγια, περί τίνος πρόκειται και με περισσότερη πραγματογνωμοσύνη, ήρθατε να επιβεβαιώσετε όλα αυτά που ε, μας απασχολούν και μας τις διάφορες επιτροπές εδώ και μήνες για να μην πω χρόνια. Πράγματα τα οποία υποπτευόμαστε, αναλύουμε, υποψιαζόμαστε και φοβούμαστε. Πάντως, τι βλέπουμε εδώ. Ότι όλες οι αιστείες κρίσης και ανάφλεξης έχουν κάποια σχέση με τις εξέλιξεις στη Ρωσία με την ρωσική πολιτική, με τους στόχους που επιδιώκει η Ρωσία. Από ό,τι φαίνεται είναι στόχος της Ρωσίας να αποσταθεροποιεί έτσι και τόσο όλες τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης αυξάνοντας ε, την εξάρτησή τους από τη Ρωσία και αφαιρώντας από την άλλη τη δυνατότητά τους να αποφασίσουν να ε, προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να τους δυσκολεύσουν να γίνουν μέλη στο ΝΑΤΟ. Άρα, από τη μια ε, αύξηση της επιρροής και από την άλλη απομόνωση ε, των χωρών αυτών για να αυξήσουν την εξάρτησή τους από τη Ρωσία. Και από την άλλη έχουμε και μια κατάσταση από τη μια έχουμε όξυνση της κατάστασης και η Ρωσία συνεισφέρει ε, για την οξύνση αυτή, αλλά από την άλλη έχουμε επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μια απόκληση ανάμεσα στην ανάλυση που κάναμε και την ε, συνειδητοποίηση της κοινή γνώμης. Και ακριβώς επειδή υπάρχει μια τέτοια απόσταση ανάμεσα ε, στην ανάλυση και τη συνειδητοποίηση της κοινή γνώμης και μέχρι και τους ηγέτες της, η Ευρώπη de facto είναι διχασμένη στη δράση αλλά και στην αντίδρασή της. Είναι αποδυναμωμένη. Οπότε, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η απόσταση και η διάσταση, έχουμε μάλλον την κατάσταση που μας προβληματίζει τι σημαίνουν όλα αυτά και τι λένε οι προγνώσεις. Δεν χρειάζονται άλλες προγνώσεις, μόνο πιο επικίνδυνο μπορεί να γίνει, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει πιο επικίνδυνο, μου φτάνει αυτός ο κίνδυνος. Τι μπορεί να κάνει και τι οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το ερώτημα. Τι μπορεί και τι οφείλει να κάνει. Από ό,τι φαίνεται οι κυρώσεις από μόνος τους δεν αρκούν. Οι κυρώσεις από μόνες τους δεν τροποποιούν συμπεριφορές. Και παγκοσμίω, αρκεί να σκεφτεί στη τη Βόρεια Κορέα. Όλο και περισσότερο ο καθένας κάνει ό,τι είχε σκοπό να κάνει ανεξαρτήτως κυρώσεων. Ανεξαρτήτως του τι σημαίνει και τι λένε γύρω-γύρω. Ο καθένας θέλει να ακολουθεί το δρόμο του και για περιμεχθεί το. Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς ακολουθούμε το δρόμο μας και εδώ έχουμε τεράστιο συνοθήλευμα κινδύνων. Και δεν είναι απλώς ένα θέμα πολέμου και ειρήνης. Είναι ζήτημα ποιότητας του, της παγκόσμιας τάξης μας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, διαμόρφωσης απόψεων και σχέσεων μεταξύ μας. Και σας ερωτώ, υπάρχει κάποια δυνατότητα αφενός χωρίς να ρίξουμε ελάδι στη φωτιά. Υπάρχει καμιά δυνατότητα αφενός να σταθεροποιήσουμε τις χώρες αυτές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από την άλλη να βοηθήσουμε να αλλάξει τακτική η Ρωσία. Γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε βρει αυτό το κλειδί και ανησυχώ. Και οι επιτυχίες της Ρωσίας στην αποσταθεροποίηση δυστυχώς αυξάνονται στις χώρες γύρω-γύρω αλλά και στην Ευρώπη και μας καθιστούν όλο και πιο αδύναμους. Περισσότερο από ό,τι θα οφείλαμε να είμαστε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ξέχασα τον Αντιπρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, τον κύριο Τιμπορζάνιεφ. Έχετε το λόγο. Αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί πραγματικά ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τους προσκεκλημένους και τους ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που διοργανώσατε αυτήν την ε, ακρόαση. Εκ μέρους λοιπόν της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την υποεπιτροπή μας για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε. Είναι με μεγάλο ενδιαφέρον που παρακολουθούμε τις εξελίξεις και με μεγάλη ανησυχία επίσης στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία και στην περιοχή του Ντόνμπας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί συνεχώς με τους συνομιλητές μας. Ένας από τους στόχους μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το ζήτημα της ασφάλειας εντός της Ουκρανίας δεν θα εξαφανιστεί από τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να ενημερώσουμε και να αυξηθεί η πληροφόρηση των πολιτών για το θέμα αυτό. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις πέρα από αυτές που ακούσαμε και από τα όσα μας είπατε. Και να πω επίσης ότι από τις παρουσιάσεις σας έλαβα κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις μου, δηλαδή την ε, αδυναμία του στρατιωτικού τομέα ε, στην Ουκρανία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, απάντησαν λοιπόν στα ερωτήματά μου και επίσης ε, τα όσα μας είπατε για την Ευρωπαϊκή Διάσταση Ασφάλειας στην Κρυμαία. Αυτά όμως είναι τα ερωτήματά μου. Καταρχάς, ίσως ο κύριος Ντεβίν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μπορούσε να μας πει περισσότερα για, την, ε, για τις σχέσεις με την Ουκρανία στον χώρο της ασφάλειας, για τις συμφωνίες μεταξύ των δύο, τη συμφωνία σύνδεσης που τέθησε ισχύ την περασμένη Παρασκευή και τις διατάξεις που υπάρχουν εκεί για ενισχυμένη συνεργασία στη, στον χώρο της ασφάλειας. Πόσο γρήγορα μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και πόσο γρήγορα μπορούμε να αναμένουμε αποτελέσματα. Μετά, η δεύτερη ερώτηση που έχω έχει να κάνει με τους ε, ανθρωπιστικούς απεσταλμένους στον Τόνμπας. Έχουμε ε, και κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις αυτοκινητοπομπές εκεί. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το τι συμβαίνει, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες και ποια στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το λόγο και αναμένω τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως η Κλέρ Μούντι με την ε, ιδιότητά της ως ε, αντιπρόεδρου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια νωρίτερα. Πράγματι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, γεμάτες πληροφορίες. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στις στοιχείες της ε, ασφάλειας στην Ανατολική Γειτονία. Από αυτά που μας είπατε, θα ήθελα καταρχάς ε, να μάθω περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις, τις βασικές υποδομές, τις ε, επιθέσεις που γίνονται, συνεχίζονται. Δεν είναι μόνο στρατιωτική η δραστηριότητα, υπάρχουν και διάφορες δράσεις που γίνονται στον κυβερνοχώρο. Και συνεχίζοντας από αυτά που είπε ένα συνάδελφος, νομίζω πως πρέπει να αποτελέσουν και αυτές οι επιθέσεις μέρος του δημόσιου διαλόγου. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με θετικά αποτελέσματα. Μετά, ε, θα σταθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σέρ για την διαφορετική οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Ρωσίας σε ό,τι αφορά την ανατολική γειτονία. Όπως είπατε κι εσείς, είναι βαθιά ριζωμένη αυτή η διαφορετική θέαση της πραγματικότητας από τη Ρωσία και αυτό που προτείνατε ως πιθανή δράση είναι να το αποδεχτούμε ή να το αναπτύξουμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, όπως ε, ακούσαμε και από αυτά που μας είπατε, να τα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, πολλά συμπεράσματα μπορούμε να αντιλήσουμε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον Ότμαν Κάρας και την ανάλυση του. Είναι πράγματι πρόβλημα ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι ένας εταίρος αδύναμος οικονομικά, πολιτικά και δυνατός μόνο στρατιωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Ρωσία μόνο στρατιωτικά είναι δυνατή, σε, καμή, σε κανέναν άλλον τομέα δεν είναι ελκυστική. Και θεωρεί όμως ότι η επιρροή της μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω απειλών, μέσω υβριδικού πολέμου, μέσω ε, εχθροπραξιών. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στον ψυχρό πόλεμο και τώρα. Μιλάμε, αν θέλετε, για παλιό καλό καιρό εντός εισαγωγικών. Στη Ρωσία αυτή τη στιγμή υπάρχουν επεκτατικές τάσεις οι οποίες ε, έχουν πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις για τους ε, γειτονές τους. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις για πόσο καιρό θα μπορέσει η Ρωσία να αντέξει το υψηλό κόστος αυτών των ε, επιχειρήσεων, αυτής της πολιτικής, για πόσο καιρό θα μπορεί να αντέξει το κόστος της κατοχής της Κρυμαίας το οποίο είναι πολύ υψηλό. Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης λοιπόν των ε, εχθροπραξιών στην Ανατολική Ουκρανία. Ε, μαζί ήμασταν στην ε, Γεωργία, είδαμε τι έγινε του στα εδάφη αυτά, είδαμε τις υποδομές, όλα αυτά κοστίζουν μεγάλα ποσά. Και όχι μόνο αυτά. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου έχει ως εξή. Ποιε είναι οι δικές σας εκτιμήσεις για πόσο μπορεί ακόμα η Ρωσία να αντέξει οικονομικά αυτό το βάρος. Και μια άλλη ερώτηση, η οποία είναι πολύ επίκαιρη νομίζω, ιδιαίτερα στα πλαίσια της άσκησης Ζάπαντ. Μας είπατε πως ο αριθμός των ε, στρατιωτών που συμμετέχουν είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, ε, εάν υπερβούν αυτόν τον αριθμό, να καλέσουν παρατηρητές. Ποια είναι τα τελευταία ε, στοιχεία που έχετε. Θα υπάρξουν παρατηρητές από το ΝΑΤΟ ή από αλλού. Θα τους γίνει πρόσκληση για να συνοδεύσουν τις ασκήσεις αυτές. Ήμασταν τον Ιούλιο με την αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία, ήταν και ε, Εξωτερικών εκεί και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να μας κατευνάσει, να μας καθησυχάσει μάλλον, να μας πει πως όλα θα πάνε καλά. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι θα αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα μετά το τέλος της άσκησης ή με την αφορμή αυτή τη άσκηση, θα αφήσουν πίσω τους διάφορες υποδομέ τις οποίες θα μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Και θα παραμείνει λοιπόν ε, ο στρατός ως παρουσία στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Λυπάμαι πάρα πολύ, θα χρειαστεί να φύγω. Αλλά θα μου διαβιβάσουν τις απαντήσεις σας. Ε, δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ε, καθηγητά κύριε Σέρ, θα μπορούσατε λίγο να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τη δική μας εξάρτηση από τη Ρωσία. Ε, ως προς τα ενεργειακά ερωτώ, κρίσιμο ερώτημα, και ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε σε μεγάλα έργα όπως είναι το North Stream. Και η δεύτερη ερώτηση, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Ντεβίνιε για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος. Το θέμα δεν το βλέπω μόνο ως δική μας αυτό άμυνα και ανθεκτικότητα δική μας, αλλά και ως δυνατότητα να αντιδράσουμε πολιτικά για, για να μην είμαστε εχμάλωτοι και όμοιροι και συνένοχοι. Γιατί αυτό είμαστε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς ξεπλένουν χρήματα Ρώσοι, Ουκρανοί και πάει λέγοντας. Και εμείς παρόλα αυτά δεν αντιδρούμε για την ανάκτηση αυτών των ε, στοιχείων. Και οι κυβερνήσει μας και τα συστήματά μας, επειδή γίνονται επενδύσει στις χώρες μας, είναι συνένοχοι. Ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία. Συμφωνείτε με αυτό που λέγουν πολλοί ότι έχει μεγάλη σχέση αυτό που κάνει ο Πούτιν για να ε, αποφύγει τις κυρώσεις Μαγνίσκη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα έγγραφα ε, του Παναμά και τη ρωσική μαφία. Και ο ε, Ξαβιενάρτ έχει υποχρέωση και θα πρέπει να φύγει. Του δίνω το λόγο, αλλά μετά πάρει το λόγο ο κύριος Σαφόζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ρωσία κατάφορα παραβίασε τη συμφωνία και της Βουδαπέστης και του Ελσίνκη. Η δημοκρατία στη Ρωσία προφανώς ε, χωράει βελτίωση και μεγάλη. Στη συνέχεια, συμφωνώ και εγώ να έχουμε μια ε, σαφή, στεναρή και κατηγορηματική θέση ως, από Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχω πάψει να πιστεύω εδώ και καιρό σε άξονες του καλού και άξονες του κακού. Επιτρέψτε μου μερικές σκέψεις. Πρώτον, όταν... Ε, ε, ανεξαρτοποιήθηκαν η Αρμενία και η Γεωργία, οι περιφερειακές συνελεύσεις της, του Ναγκόρνου Καραμπάχ και της Νότιας Οσετίας δεν δέχτηκαν να ενταχθούν ε, στις επικράτειες που τους είχαν κατατάξει στη Σοβιετική εποχή. Τότε είχαμε ε, με τα κριτήρια του Μίνσκ συμφωνίες στη Μαδρίτ και μιλούσαμε για αυτοδιάθεση στο Νο Καραμπάχ. Πού είναι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το πολιτικό κριτήριο που σημαίνει ε, ότι σπάμε την εδαφική ακαιρεότητα για να δώσουμε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση στο Όριο Καραμπάχ, στο Ορεινό Καραμπάχ και γιατί για την Νότια αιτία αυτό μας φαίνεται κακό. Δεν είναι αυτό το κουτί της Πανδώρας που θα καταλήξει στην Κρυμαία. δεν έχουν όλοι το ίδιο λόμπι όπως έχει η Αρμενία στη Γαλλία και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Μήπως αυτή είναι η διαφορά, γιατί κατά τα άλλα είναι όλα ίδια. Το 1940 ε, ε, έγινε μια εισβολή της Γερμανίας ε, που εισέβαλε ε, στο Βέλγιο και στη Γαλλία και δεν είδα κανένα Βέλγο και κανένα Γάλλο να φεύγουν προς τη Γερμανία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε εκατοντάδε. χιλιάδες κόσμο που προσπαθεί να καταφύγει, να βρει ε, προστασία στη Ρωσία. Άρα κάτι γίνεται εκεί. Όταν ακούω ότι, ότι δεν είναι φίλια σύραξη, είναι σαν να λέμε ότι στην Συρία δεν είναι φίλια σύραξη. Και βεβαίως υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει. Αλίμονο. Και για τους πρόσφυγες. Κάποιο είπε ότι πρόσφυγε είναι ένα δημοψήφισμα που γίνεται με τα πόδια, ότι πηγαίνει στη διπλανή χώρα. Και περίπου 10% του πληθυσμού της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή ζει στη Ρωσία και δεν αισθάνεται ε, ότι η Ρωσία είναι μια εχθρική χώρα. Εγώ είμαι δικηγόρος και έχω ζήσει τον νόμο και την νομιμότητα επί Φράγκο. Ο νόμος είναι τύπος, δεν είναι πραγματικότητα. Άρα ένα καθεστώς απολύτως διεφθαρμένο, με τελευταίο παράδειγμα η αφαίρεση της ηθαγένειας του Σαχασβίλη, που δεν είναι και καμιά Παναγίτσα κι αυτός, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ολιγάρχες που αλωνίζουν και βλέπουμε ότι στη Μολδαβία κερδίζουν εκείνοι που είναι υπέρ των Ρώσων. Προφανώς γιατί βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους διεφθαρμένους. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις ε, νομιμότητες και να περάσουμε στις πραγματικότητες. Και ε, στην Ουκρανία ε, οργίαζε η διαφθορά. Και εκεί είναι η άμυνα και η ανθεκτικότητα και το ηθικό της κοινωνίας. Ούτε τάγκς, ούτε άρματα μάχης, ούτε συστοιχίες, ούτε τίποτα. Μας εκπλήσει που θέλει η Ρωσία να έχει μια σφαίρα επιρροής και σας ερωτώ, δεν έχουν οι δεν έχει η Κίνα, γιατί παραμένουν στην Κορέα γιατί η Κίνα έχει συμφέροντα στη Βόρεια Κορέα και εισέβαλαν στη Γρανάδα Ηνωμένε Πολιτείε για συμφέροντα του Παναμά. Οι υπερδυνάμεις συμφέροντα έχουν. Είναι πραγματικά συμφέροντα και η πραγματικότητα και η πολιτική γίνεται με πραγματικότητες και η φιλολογία και η φιλοσοφία είναι γυαλού. Αν δείτε τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μείνετε εμβρόντιτοι. Κατά πλειοψηφία εγκρίναμε ένα ψήφισμα για τη Μαύρη Θάλασσα που έλεγε ότι στηρίζαμε ε, άξονα στρατιωτικής συνεργασίας Μολδαβίας, Ουκρανίας, Γεωργίας. Αυτό σας φαίνεται ρεαλιστική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο ίδιο ψήφισμα να λέμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ηγεμονία μας στον εύξηνο πόντο. Όταν εισέβαλε, γιατί εισέβαλε στην Κρυμαία παράνομα, παράνομα Ήρθα σε επαφή ε, με τον στρατιωτικό ακόλουθο της ε, Τουρκίας, της τουρκικής πρεσβείας και τους λέω έχετε προβλέψει την ρωσική στρατιωτική παρουσία ε, της Ρωσίας στην Κρυμαία. Μου λέει όχι, δεν αλλάζουμε δόγμα. Άρα ο βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην περιοχή δεν θεωρείται ότι απειλείται. Μένω έκπληκτος με αυτά που ακούω πυρηνικό πόλεμο δηλαδή φοβάστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταστραφούν οι πάντες συμπεριλαμβανομένε τη Ρωσία. Σας φαίνεται περίεργο ότι έχει συμφέροντα στη Συρία. Αν δείτε το χάρτη, η Συρία είναι πιο κοντά στη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γιατί έχει πάει εκεί, γιατί εμείς είμαστε αδρανείς ε, όλα αυτά τα χρόνια και δεν καταφέραμε να στηρίξουμε αυτό που θα έπρεπε, που είναι ελεύθερος Συριακός στρατός. Συμπέρασμα και που καταλήξαμε στους ε, Ισλαμιστές, ε, τους Σαουδάραβες Ουαχαμπίτες. Βεβαίως έχει συμφέροντα εκεί, γιατί και οι τζιχαντιστές επιστρέφουν στη Ρωσία. Θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Ε, να ολοκληρώνεται, λέει η πρόεδρο. Ναι, ναι, τελειώνω, πρόεδρε. Αν δεν είμαστε ε, σε θέση να καταλάβουμε ποιο είναι ο αντίπαλό μα, θα δημιουργήσουμε ένα δογματικό δόγμα και, ε, που δεν θα μα οδηγήσει πουθενά. Mr. Schaffhauser. Ο κύριος Σαφοζέρ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Άκουσα με χαρά τον συνάδελφο Νάχτο, ο οποίος λέει ε, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επιθετικός, ενώ εγώ θα είμαι, κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι δεδομένα. Να υπενθυμίσω επίσης τον κύριο Καράς ότι ευτυχώς που έχουμε και τα Υπουργεία Εξωτερικών, ευτυχώ που έχουμε τα κράτη που είναι καλύτερα πληροφορημένα από αυτό το κοινοβούλιο, που έχουν την αίσθηση της ιστορικότητας ε, του πολιτισμού και πρέπει να διαχειριστούν πραγματικά τις διεθνείς σχέσεις, όχι σαν και εμάς, γιατί αν πραγματικά ακούγαμε το τι θέλει το Κοινοβούλιο για τη Ρωσία στην εξωτερική πολιτική, προφανώς θα προετοιμάζαμε ένα πυρηνικό πόλεμο όπως το υπογράμμισε και ο Νάρτ. Ευτυχώς που έχουμε χώρες σαν την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία που δεν συμφωνούν με το Κοινοβούλιο γιατί αλλιώς δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν. Να πω επίσης στην κυρία Φώτιγκα ότι είναι κρίμα που πολωνοποιούμε ουσιαστικά την εξωτερική μας πολιτική. Γνωρίζω την Πολωνία, είναι μια φίλη χώρα, έχω πάει αρκετές φορές και θα ήθελα να πω ότι και στην Πολωνία δεν υπάρχει μια τόσο, θα έλεγα, απόλυτη θέση καρικατούρα σε σχέση με τη Ρωσία. Θυμάμαι κάποιους φίλους που μου έλεγαν ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, μεταξύ των οποίων και τον μακαριστό Ιωάννη Παύλο. Να πω επίσης ε, ότι πρέπει να θυμίσω ότι ορισμένα θέματα ε, απαιτούν να δοθούν απαντήσεις. Κύριε Σάρ, είπατε ότι υπάρχουν ζώνες επιρροής. Όπως είπε επίσης ο συνάδελφος Ναρτ, ποια είναι η χώρα, ποια είναι η ισχυρή δύναμη που δεν έχει ζώνες επιρροής. Γι' αυτό εκπλήσωμε ε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματική η Ρωσία. Αν βλέπουμε τη ζώνη επιρροή της το 89 με την πτώση του τείχους και η ιδέα τότε υποτίθεται ήταν να παραμείνουμε στις ισορροπίες της εποχής και δούμε το τι συμβαίνει σήμερα με το ΝΑΤΟ σαν παράδειγμα βλέπουμε ότι έχει υπάρξει έλλειψη επιρροής και πτώση κυριαρχίας της Ρωσίας. Λοιπόν, τι θέτε θέμα αποτελεσματικότητας της πολιτικής της Ρωσίας. Ποιοι είναι επιθετικοί, οι Ρώσοι ή οι δυτικές δυνάμεις, βλέποντας ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αναφέρεστε και στη σχέση με το Γιαννούκοβιτς το 2013. Γιατί αν ο Γιαννούκοβιτς ήθελε μια ισορροπημένη πολιτική και σωστά το υπογραμμίσατε, γιατί έγινε το πραξικόπημα ενώ το Φεβρουάριο είχαν καταλήξει στις συμφωνίες για να ισχύσουν το 2014. Γιατί έγινε λοιπόν αυτό το πραξικόπημα και γιατί ο Γιαννούκοβιτς προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του και την ίδια του τη ζωή άλλωστε ζητώντας την προστασία των Ρώσων. Μια και έχετε μια μακρόπρόθεσμη πολιτική ε, αντίληψη για την ιστορία, να υπογραμμίσετε το πώς η Ρωσία θέλησε να παίξει με την πολιτική ε, του ΝΑΤΟ. Θυμηθείτε τις προσπάθειες του Ρογκώση. Γιατί δεν πέτυχε αυτό. Τίθενται όλα αυτά τα θέματα. Λέτε ότι η CIA και οι αντικατασκοπίες και κάποιες άλλες απόψεις από τον ε, Αμερικανό Πρόεδρο υπογραμμίζεται αυτό το οποίο έλεγε ο Ρούσβελτ, ότι υπάρχει δηλαδή ε, το σύνολο γενικά ο μηχανισμός στρατιωτικής βιομηχανίας και στρατού φυσικά που θέλει να διοικεί τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, βγάλτε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ο πρόεδρος είχε υπογραμμίσει μία αλφα πολιτική και τώρα ακολουθείται μία β και όταν λέμε ότι η Ρωσία πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη, γιατί αλλάζει στο εσωτερικό της λόγω της Ρωσίας ή λόγω των ειδικών της εσωτερικών αντιθέσεων και λόγω της άρνησης να δει την πραγματικότητα. Παρακαλώ να ζητήσω και από εσάς κύριε Σαφοζέρ να τελειώνετε. Κοιτάξτε, πρόεδρε, συγγνώμη, είναι θέματα όπως ε, τα έθεσε και ο κύριος Καράς, μπόρεσε το χρόνο, είχε το χρόνο, γι' αυτό πραγματικά ισορροπήστε λίγο τον χρόνο. Εγώ είμαι ένας από τους λίγους που έχουν αντίθετη άποψη και όμως αντιπροσωπεύω το 40 και το 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, Τελειώνω, τελειώνω λέει ο κύριος Σαφοζέ, τελειώνω. Συνάδελφοι, μπορείτε να επιτρέψετε στον κύριο Σαφάουζερ να ολοκληρώσει. Για τον κύριο Ράτς, θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμίσουμε το τι έγινε στη Γεωργία. Η γαλλική κυβέρνηση με είχε στείλει στη Γεωργία το 2008. Ποιος ήταν υπεύθυνο ο Σακασβίλη, με τη CIA ή μήπως οι Ρώσοι. Ποιοι ήταν αυτοί που οδήγησαν στη σύγκρουση στη Γεωργία. Η Γαλλία έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση γύρω από το θέμα αυτό. Στην Ουκρανία το ίδιο, ίσως θα είναι χρήσιμο. Να ξαναδείτε το τι έγινε στις 21 και 22 Φεβρουαρίου πριν μιλήσετε για την προσάρτηση της Κρυμαίας να δείτε τι συνέβη και τότε θα μπορέσουμε να δούμε και για τη Συρία. Ποιος αποσταθεροποίησε τον Ασάντ, ποιος ε, αυτή τη στιγμή συμμάχησε με τους τζιχαντιστές, οι δικές μας δημοκρατικές χώρες και το παραδέχονται σήμερα. Ο Γάλλος Πρόεδρος παραδέχεται ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική, γιατί η πολιτική που ακολουθούμε δεν είναι η πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, αλλά η πολιτική των λόμπι που εκπροσωπούν τις στρατιωτικές και βιομηχανικές αμερικανικές δυνάμεις εναντίον της δημοκρατίας που αποφελούνται από τα εγκλήματα. Κύριε Σαφοζέρ παρακαλώ τελειώνετε. Λοιπόν, είναι δύσκολο να έχει κανείς αντίθετη άποψη μέσα σε αυτή την Επιτροπή, γιατί η πραγματικότητα και η ιστορία δυστυχώς δεν γίνονται αποδεκτές. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν φανταζόμουν ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα οι υποστηριχτές της Ρωσίας θα ακουγόντουσαν τόσο δυνατά και θα ήταν τόσο πολλοί παρόντες. Είναι πραγματικός λόγος ανησυχίας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν μαθήματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πώς να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Ας ε, μας προστατεύσει ο Θεός από τους φίλους απέναντι στους εχθρούς. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Σαφοζέ. Δεν σας διακόψαμε. Λοιπόν, έχω να θέσω δύο ή τρεις ερωτήσεις, λέει ο κύριος Μποστινάρο. Πώς παρουσιάζεται η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς ενισχύεται ο συντονισμός με τις Ηνωμένε Πολιτείες απέναντι στην ρωσική απειλή και επιθετικότητα, γνωρίζοντας ότι μόνες μας καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι μπορεί να επικρατήσει. Και γνωρίζοντας επίσης ότι ο οι διάφοροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγουν ότι ο Πουτίν δεν είναι εχθρός αλλά εταίρος. Οπότε διαρωτώ με εδώ τι σημαίνει εταίρος σε μια περίοδο απειλών για την ασφάλεια. Δεύτερη ερώτηση. Τι ρόλο θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αυτό συζητάμε και θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι ικανή να καλύψει κάποιες από τις ανάγκες της στον τομέα της ασφάλειας γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες διεθνούς ασφαλείας έχουν αλλάξει και η απειλή στην Ανατολική Ευρώπη είναι βασικό εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ενότητα. Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω επίσης ε, ε, ένα σοβιετικό κινηματογραφικό έργο το οποίο είχε τίτλο «Η Μόσχα δεν πιστεύει στα δάκρυα, ούτε κι εγώ». Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να αναπτυχθεί θεωρώντας ότι η Ρωσία είναι σεβαστός εταίρος. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τις αξίες της και τα σύνορά της και τότε μόνο θα τη η Ρωσία. Μπορούμε να προστατεύσουμε, λέγανε οι Λατίνοι, ή συγγνώμη οι Ρωμαίοι, ε, την ειρήνη ετοιμαζόμενη, προετοιμαζόμενη για τον πόλεμο. Έτσι μόνο θα διασώσουμε την ε, ενότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριος Γιούρεκ. Γίνεται λόγος λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δύναμη που πρέπει να χρησιμοποιήσει soft power, ήπια δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε και τι γίνεται στις χώρες αυτές, τι γίνεται με τα κόμματα της Ουκρανίας και τι γίνεται με τις πολιτικές δυνάμεις εδώ. Έχουμε δει, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας ε, πολωνός ευρωβουλευτής, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα με την Ουκρανία. Έλαβε τέλος, βέβαια, αυτό το θέμα. Μετά μην ξεχνάμε πως υπάρχει μία μικρή καθολική μειονότητα στην Ουκρανία. Έχουν, μάλιστα, και καρδινάλιο. Εκλέγουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε όλες αυτές τις πτυχές. Η Ουκρανία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, με πολλές πτυχές. Μια χώρα στην οποία σίγουρα μπορούμε να δώσουμε ε, διάφορες, ε, διάφορα πράγματα να κάνει, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια κυρίαρχη χώρα με έδαφος. Επίσης υπάρχουν πολλές ε, και διαφορετικές απόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την Νότια Οσετία, αλλά το θέμα είναι να βρούμε μία ειρηνική λύση για να δοθεί ένα τέλος στις διαμάχες. Στην Ουκρανία πιστεύω πως το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από την άλλη, από τις αρχές της ε, δεκαετίας του 50 υπάρχει μία φυσική απειλή μια πληθυσμιακής ομάδας. Στην ε, Ανατολία το είδαμε πριν από έναν αιώνα αυτό, όμως ε, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ πιο πρόσφατα. Εάν θέλουμε λοιπόν να λύσουμε τα προβλήματα, τότε πρέπει να εξετάσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γιατί έχει η κάθε περίπτωση τις δικές της ιδιαιτερότητες και να γνωρίζουμε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάμε. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουμε και εταίρους στην εξωτερική μας πολιτική. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις χώρες αυτές ως απικίες, αλλά ως εταίρους. Ίσους εταίρους που έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτά λοιπόν τα δικά μου συμπεράσματα στα όσα άκουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας με αντίστροφη σειρά, αρχίζοντας με, από την Μαρία Ντούνερ. Δυστυχώς δεν υπάρχει πολύς χρόνος για απαντήσεις. Στις πολλές ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Δεν θα σας δώσω ε, χρονικό περιθώριο, όμως σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα πολεμικά, η κυρία Ντίνερ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση του κυρίου Σντρογεύσκη για τις προγνώσεις σχετικά με την κατάσταση. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε κληθεί να κάνουμε στο Ινστιτούτο μας. Να δώσουμε απαντήσεις και αξιόπιστες προγνώσεις. Προσπαθούμε όμως να παρακολουθήσουμε με προσοχή την κατάσταση, να εξετάσουμε και να επαληθεύσουμε ε, την κάθε μας πηγή και να μην μας ξεφεύγουν λεπτομέρειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρυμαία, ναι, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες ε, προβλέψεις, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Ποια δηλαδή θα πρέπει να είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, πράξεις της Ρωσίας. Θα έπρεπε να είναι στρατιωτική απάντηση, αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το ΝΑΤΟ όμως είναι ο αρμόδιος οργανισμός εδώ έχει τα μέσα, έχει την αρμοδιότητα έτσι ώστε η Ρωσία να μην έχει την εντύπωση πως καθυστερούμε, πως χρονοτριβούμε, πως ε, αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι και ο αρμόδιος ε, οργανισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια τη Ρωσία και τους στόχους της, υπάρχουν διασυνδέσεις, υπάρχει μια ήπια δύναμη ε, που προσπαθεί να ασκήσει η Ρωσία σε συνδυασμό με την σκληρή στάση Τώρα, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στις ε, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Φοβάμαι πως όχι. Όχι, δυστυχώς, διότι, όπως φάνηκε, η Ρωσία έχει διαφορετική αντίληψη για τον μετασοβιετικό χώρο από ότι Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες χώρες και αυτό έχει και συγκεκριμένες συνέπειες για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Πρώτον, ε, θεωρώ πως πρέπει να έχουν την ε, δυνατότητα αυτές οι χώρες να κάνουν ελεύθερες εκλογές και δεύτερον, εμείς να τις στηρίξουμε. Πώς όμως μπορούμε να τις στηρίξουμε έτσι ώστε η Ρωσία να μην παρεμβαίνει με τρόπο που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Μία δυνατότητα σίγουρα είναι η στρατιωτική επέμβαση. Ίσως ε, ένας ε, Πολωνός φίλος από το Υπουργείο Εξωτερικών ε, είδε ο ίδιος με τα μάτια του την κατάσταση και μας είπε πως ο στρατός πολλές φορές δεν έχει κράνη, δεν έχει την κατάλληλη εξάρτηση. υπάρχουν πολλά προβλήματα, πρακτικά προβλήματα, καθημερινά. Τώρα, για πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει η Ρωσία τον πόλεμο στην Κρυμαία. Να το πούμε αλλιώ ίσως. Η Κρυμαία έχει οχυρωθεί, έχει γίνει ένα πολύ καλά οχυρωμένο φρούριο. Η Ρωσία δεν υπολογίζει χρήματα, προσπαθεί να οχυρώσει όσο, το καλύτερο, όσο πιο καλά μπορεί την Κρυμαία. Πρέπει να πάμε λοιπόν ε, στην πηγή. Δεν έχω αξιόπιστες πηγές λοιπόν για το ποσό, όμως σίγουρα είναι πολύ ψηλό. Μπορούμε όμως να εξετάσουμε και άλλες πτυχές, ε, κοινωνικές πτυχές. Ε, για παράδειγμα, στην Κρυμαία υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Το συνταξιοδοτικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα. γιατί τι συντάξεις είναι υπεύθυνη η Ρωσία και όχι η Ουκρανία. Λευκορωσία τώρα, αποστολή παρατηρητών στην άσκηση. Ναι, Ζητήσαμε 12 παρατηρητές υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, όμως υπάρχουν άλλοι κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή τους. Και μάλλον για τη Λευκορωσία είναι κάποιες εγγυήσεις η συμμετοχή αυτών των παρατηρητών απέναντι στη Ρωσία. Νομίζω όμως πως η Ρωσία θα αποσύρει τα στρατεύματά της μετά το τέλος της άσκησης. είτε μετά από παράκληση της ίδιας της ε, Λευκορωσίας. Επίσης υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα πυραυλικά συστήματα Λευκορωσία και Ρωσία. Ε, τώρα, μία ξεκάθαρη στάση ενωμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Αυτό είναι δύσκολο. Είναι όμως πολύ καλό να απαντούμε ενωμένα και να μην εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση διχασμένη, είτε όταν πρόκειται για κυρώσεις είτε για κάποια άλλη αντίδραση. Ε, προσπαθούν βέβαια να διχάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε να συμβεί αυτό. Και όπως είπα, εδώ είστε εσείς στο επίκεντρο. Έχετε πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις σας. Ο καθηγητής κ. ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Με αντίστροφη σειρά όπως πρότεινε και η Πρόεδρος. Λοιπόν, θα προσπαθήσω πρώτα απ' όλα να απαντήσω την ερώτηση που μου απίφθηνε ο κύριος Σάφοζερ. Συμφωνώ πάρα πολύ ε, να ασχολούμαστε με τα γεγονότα. Έχουν μεγάλη σημασία τα γεγονότα. Το Φεβρουάριο 2014 ήταν πλήρως νομιμοποιημένη αλλαγή εξουσίας. Όχι. Το Σύνταγμα ε, προβλέπει πώς καθαιρείται ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Γιαννουκόβιτς δεν καθαιρέθηκε με βάση τη διαδικασία. Ωστόσο, από το Μάιο του 2014 έχει πρόεδρο η χώρα και από τον Οκτώβριο του 2014 κοινοβούλιο και κυβέρνηση με πλήρη νομιμοποίηση. Η νομιμοποίηση των Ουκρανικών αρχών ε, είναι δεδομένη γιατί έχουν εκλεγεί με τις πιο καθαρές εκλογές που είχε ποτέ η Ουκρανία. Η νομιμοποίηση τους λοιπόν και του Προέδρου και της κυβέρνησης και της Βουλής είναι κάτι που αναγνωρίζει και η Ρωσία. Για να έρθω και πάλι σε γεγονότα. Υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο κύριος Γιανουκόβιτς ε, φώναξε τους Ρώσους για να ε, σωθεί ο ίδιος. Και πάλι να δούμε τι έγινε. Τα γεγονότα σύμφωνα με ε, το σύνταγμα της χώρας, ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα μόνος του να προσκαλέσει ξένα στρατεύματα στη χώρα. Αυτά για τα γεγονότα. Απαντώ στον κύριο Γκάλε για το πώς μπορεί η Ρωσία να διατηρεί σε προσάρτηση την Κρυμαία και την παρουσία της ε, στην κοιλάδα του Ντόν, στον Ντόμπας. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η Κρυμαία, σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο, είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν πρόκειται ποτέ να την εγκαταλείψει η ε, Ρωσία. Βεβαίως επιβαρύνει πολύ ε, τον προπολογισμό. Δύο εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι της Κρυμαίας, πολλά πεινασμένα στόματα να ταΐσεις. Θα κάνει ό,τι μπορεί όμως η Ρωσία για να διατηρήσει ε, την Κρυμαία και σε λειτουργία. Θα ολοκληρωθεί ε, προσεχώς και μια γέφυρα ε, που θα βοηθήσει πολύ τον προπολογισμό. Για την περιοχή του Ντόνμπα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι το κόστος, ούτε μέχρι πότε μπορούν να αντέξουν. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι ανησυχούν για το κόστος εκεί στην Ουκρανία. Και αυτό επίσης εξηγεί για ποιο λόγο η Ρωσία θα προτιμούσε να επανέλθει η περιφέρεια αυτή στην Ουκρανία, αλλά με τους όρους της Ρωσίας. Γιατί το λογαριασμό θα τον πληρώσει η Ουκρανία τελικά. Απαντώ στον κύριο Σάνη για ε, τις ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές στην αρχή ήταν μεγάλη η αδιαφάνεια για το τι μετέφεραν εκεί. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι είναι πραγματικά ανθρωπιστική βοήθεια αυτή που μεταφέρεται εκεί. 65 τέτοιες αυτοκινητοπομπές. Οι περισσότερες έχουν περάσει στην Ανατολική ε, Ουκρανία ε, φυλάκια του ΟΑΣΕ που κάνει ελέγχους. Αν θέλει η Ρωσία να βάλει κάτι στην Ουκρανία ή να βγάλει κάτι από την Ουκρανία, δεν χρειάζεται να περάσει από επίσημους μεθοριακούς σταθμούς ε, που ελέγχει ο ΟΑΣΕ ή επίσημες αυτοκινητοπομπές. Μπορούν να περάσουν όποτε θέλουν από τα σύνορα ό,τι θέλουν. Και για την ενημέρωσή σας υπάρχουν πολλά βίντεο, μαγνητοφωνήσεις κτλ. Όταν ξεφορτώνουν τα φορτηγά αυτό που κατεβάζουν ανθρωπιστική βοήθεια παίζουν σημαντικό ρόλο στο να δίνουν στον εναπομείναντα πληθυσμό κάποια στοιχειώδη ε, ακριβώς ανθρωπιστική βοήθεια. Σε ό,τι αφορά το αεροπλάνο ε, που καταρρίφθηκε, ε, ε MH17, ε, ε, έχουν ομολογήσει ότι είναι λάθος. Ότι έκανε λάθος ως προς το στόχο. Είναι γνωστά ε, το, το τι όπλο χρησιμοποιήθηκε και μάλλον γνωστό και γνωστή και η ιδιότητα εκείνων που το διέπραξαν, αλλά είναι μάλλον αμφίβολο αν θα προσταχθούν στη δικαιοσύνη. τι θα κάνουμε τώρα για τις κυρώσεις. Λέτε ότι δεν επαρκούν και δεν αλλάζουν την κατάσταση. Συμφωνώ απολύτως. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ότι η άρση των κυρώσεων είναι αυτή που θα άλλαζε την κατάσταση. Γιατί σε περίπτωση που αρθούν οι κυρώσεις, οι Ρώσοι θα το ερμηνεύσουν ως πράσινο φως ότι εντάξει είχαμε λίγα χρόνια προβλήματα αλλά τώρα σε επανέλθουμε στα παλιά. Ακόμα και αν δεν βοηθούν οι κυρώσεις όπως ήταν η αρχική πρόθεση η άρση τους τώρα θα βλάψει ακόμα περισσότερο. Το πώς να επηρεάσουμε τη Ρωσία ρωτήσατε και πώς να σταθεροποιήσουμε τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Συνδέονται τα δύο αυτά ερωτήματα μεταξύ τους αν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση και το μετασχηματισμό των μετασοβιετικών χωρών, εδώ μιλώ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία κυρίως, θα ε, είναι αυτό ένα παράδειγμα και για το ρωσικό πληθυσμό. Και ο μέσος Ρώσος ψηφοφόρος θα καταλάβει ότι αφού τα κατάφεραν οι Ουκρανοί, γιατί να μην τα καταφέρουμε και εμείς οι Ρώσοι. Και στην ερώτηση του κυρίου για τις προβλέψεις, θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στην πρόγνωση μας. Ας το τολμήσω για τον Ντόμπας. Μπορεί ακόμα αρκετά χρόνια να αντέξει. Είναι μια σύραξη χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλού κόστους. Χρησιμοποιούν κάτι δεύτερα και κάτι τρίτα συστήματα οπλικά και αυτό που ε, δημιουργείται εκεί, προκαλείται μάλλον ως δεινά και ως πόνος είναι κυρίως για τον τόπιο πληθυσμό και όχι για τους Ρώσους. Ο κύριος, Ο έχει το λόγο. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω την εντυπωσιακή ακρίβεια του κυρίου Ρας. Νομίζω ότι η συμπεριφορά των Ρώσων από το 1999 και μετά ήδη από τότε στη σύγκρουση στο Κωσυφοπαίδιο και είχε χρησιμοποιηθεί υλικό διτής χρήσης. Το υλικό αυτό το είχαν αποστείλει στο Υπουργείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Υπεύθυνο τότε ήταν ο Σέργεϊ Σοϊγκού, ο οποίος σήμερα είναι Υπουργός Άμυνας. Θα συμφωνήσω λοιπόν με αυτά που είπε ο άντρας, ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το 15 ή 20% του υλικού, το οποίο δεν είναι απόλυτα συμβατό με τους κανόνες που είναι ενισχύ. Και νομίζω ότι αυτό που είναι σαφές είναι ότι το 2014 μία από τις αποστολές αυτές είχε σαν στόχο να απομακρύνει από τον πάσ τέτοιου είδους ε, υλικό. Λοιπόν τώρα θα είμαι σύντομος από εδώ και πέρα. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις ε, φυσικά θέλουν να έχουν σφαίρες επιρροής. Το θέμα είναι επί ποιας βάσεως διαμορφώνονται οι βάσεις αυτές επιρροής. Διαμορφώνονται επί τη βάση επιλογών, θα έλεγα ελεύθερων. μια χώρα θέλει να ανήκει σε μια τέτοια ζώνη ή αναγκάζεται να ανήκει σε μια τέτοια ζώνη. Νομίζω ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου κανονικά υπάρχει υπογράμμιση και μεγάλη σημασία στην ελεύθερη βούληση και την επιλογή. Κάθε χώρα πρέπει να είναι ελεύθερη να επιλέξει τις συμμαχίες της και εδώ γίνεται η διάκριση αν θέλετε. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το έθεσε ένας άλλος εξαιρετικός σας συνάδελφος για την παρούσα κρίση στην Ουκρανία. Στην περίπτωση του Ντόνμπας, όπως επίσης και σε άλλους ε, πολέμους ε, στην περιφέρεια της Ρωσίας για εκατοντάδες χρόνια, υπάρχει ένα μείγμα θα έλεγα συμμετοχής κρατικών πρωταγωνιστών, ε, παρακρατικών, εσωτερικών και εξωτερικών. Είναι γεγονός όμως ότι σε καμία περίπτωση μέχρι τώρα δεν υπήρξαν θα έλεγα σεβαστές ε, διεθνείς οργανώσεις και υπήρξαν ορισμένες ε, που έλεγαν ότι μόνο το 25% των Ουκρανών ε, θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Είπαν λοιπόν ότι το 40% και όχι παραπάνω όλων των ομπλάστ της Ουκρανίας έχουν εκφράσει την επιθυμία να συνδεθούν με τη Ρωσία και όχι με την Ουκρανία. Είναι σαφές ότι ιδιαίτερα οι αρχές των περιοχών του Λουχάνσκ και των περιοχών του Ντονμπάς ήταν περισσότεροι Ρώσοι στην καταγωγή όπως ο Γκίρκιν, ο Στερκόφ και άλλοι οι οποίοι ανήκαν στην μυστική υπηρεσία της Ρωσίας και οι οποίοι παραπονούνται γιατί δεν βρίσκουν αρκετούς να πολεμήσουν για τη ρωσική πλευρά και δυστυχώς προσφεύγουν στη χρήση φυλακισμένων κτλ. Τώρα υπάρχει το θέμα των προσφύγων. 1.700.000 είναι αυτοί που ζουν στην Ουκρανία αντίθετα με αυτούς που πήγαν στην Ρωσία. Έπρεπε να διασχίσουν μια εμπόλεμη περιοχή, μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά το έκαναν αυτό παρά τις δυσκολίες. Εδώ γνωρίζω αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ στο, στη δεκαετία του 90 και μετά είχα πάει και στο Ντονέτσκ και σε, στη Μαριούπολη και σε άλλες περιοχές και έχει σημασία να δει κανεί ε, πώς μετακινήθηκαν οι άνθρωποι και που ζουν σήμερα. Για το θέμα της διαφθοράς, ε, ίσως εδώ να εκφράσω τον εντυπωσιασμό μου. Αν μια χώρα πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά, είναι η Ουκρανία, αλλά δεν μπορεί να το ζητάει η Ρωσία αυτό. Νομίζω ότι η διαφθορά στη Ρωσία ταυτίζεται με τους κρατικούς μηχανισμούς, αντίθετα από τις άλλες χώρες. Η διαφθορά στην Ουκρανία είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταπολεμηθεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν πολιτικά κόμματα, υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ελεύθερη κοινωνία των πολιτών και όλοι εκτίθενται και πιέζονται. Και αυτά θα έλεγα εντάσσονται στη λεγόμενη μετασοβιετική τάξη. Ένα άλλο μέλος της Επιτροπής σας είπε, και το καταλαβαίνω αυτό, ότι η Ρωσία είναι στρατιωτικά ισχυρή, αλλά όχι σε άλλους τομείς. Είναι χειρότερη η κατάσταση δυστυχώς. Αυτό το οποίο έχει η Ρωσία κοινό με τις ελίτ τις διαφθαρμένες είναι θα έλεγα ένα δίκτυο δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συνδέει την εξουσία με το χρήμα και ε, θα έλεγα σε αυτό το δίκτυο υπόκεινται όλες οι περιφερειακές, τοπικές και κεντρικές αρχές. Και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό κίνητρο ε, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει οι αντιλήψεις που βασίζονται στο σεβασμό του νόμου και των δικαιωμάτων να ισχύουν στις περιφερειακές στη Ρωσία χώρες δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεσή μου. Ε, μία σύντομη ίσως απάντηση αν μου επιτρέψετε. Στη σημαντική ερώτηση της κυρίας Μούντι. Τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι δράση θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους εταίρους της Ανατολικής Γειτονίας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λογικοί και ρεαλιστές. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα να πούμε σε όλους αυτούς τους εταίρους, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι η δυνατότητα μόχλευσης επιρροής που έχουμε είναι περιορισμένη. Η Ρωσία έχει την ικανότητα και απέδειξε ότι έχει και τη βούληση, ακόμα και αν θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε, να σταματήσει τις σχέσεις αυτές. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σε μεμονωμένη φάση να έχουμε μια πραγματική συζήτηση για το τι θέλουμε να κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη στις πιέσεις που υφίσταστε. Πού μπορεί η βοήθειά μας να βοηθήσει. Νομίζω μόνο σε αυτήν την περιορισμένη αλλά και μετριοπαθή βάση θα μπορέσουμε ίσως να πετύχουμε κάτι και να ξεφύγουμε από γενικού τύπου συζητήσεις. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά νομίζω ότι η Πρόεδρος θα με επαναφέρει στην τάξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομο. Να ζητήσω από τον προτέρων συγγνώμη για το σύντομο των απαντήσεών μου στι άμεσε ερωτήσει και ευθείε ερωτήσει που έκαναν οι Ευρωβουλευτέ. Πρώτον, ε, η συνεργασία στον τομέα τη ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία. Ναι, υπάρχει τέτοια διάταξη στην Συμφωνία Σύνδεση υπάρχουν συνεχιζόμενες δράσεις, ε, θετικές οι τάσεις. Υπάρχει η αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία, στην οποία περιέχονται συγκεκριμένες ε, καθευθυντήριες γραμμές και καθοδήγηση για ε, τα θέματα αυτά στα πλαίσια της, των αποστολών της ε, πολιτικής, κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Μετά υπάρχουν διάφορες συναντήσεις που γίνονται εδώ και καιρό για τα θέματα αυτό, ε, αυτά. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκόμες για την διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματο, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά να τονίσω και πάλι εδώ ότι αυτό που κάνουμε εμείς στην Ουκρανία έχει αποφέρει αποτέλεσμα, έχουμε δει πρόοδο. αρχίζει να δημιουργείται ένα σύστημα διαφάνειας το οποίο ε, στην Ουκρανία φτάνει πέρα από αυτά που έχουν ζητηθεί. Ξεπερνά μάλιστα και το σύστημα διαφάνειας ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, δράσεις που γίνονται. Η εισαγγελία έχει ε, δράση. Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα πληστηριασμών, ένα καινούργιο σύστημα το οποίο είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Παραμένει σίγουρα διαφθορά στην Ουκρανία. Είναι και αυτή ανθεκτική όπως και η χώρα σε άλλα θέματα. Και φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε η Ουκρανία να καλύψει 25 χρόνια διαφθοράς μέσα σε λίγους μήνες. Τώρα, ο κύριος ε, Σεφχάουζερ έκανε μια ερώτηση, την οποία θα απαντήσω στα γαλλικά. Έχει διερμηνία άλλωστε. Μιλήσατε για την πολωνοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό θα άρεσε στην Πρόεδρο, γιατί ε, ε περιπεί μεγάλη τιμή στην Πολωνία Βέβαια μεγάλη χώρα με 40 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά λέμε ότι επιβάλλει και την πολιτική σε 500 εκατομμύρια. Ε, για να σοβαρευτούμε λίγο, η πολιτική ανατολική γειτονία. Ε, ο Σύνοδος Κορυφής της Ρήγας, ο Βίλνιους και η αποφάση για τη Ρωσία επάρτησαν ομόφωνα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Έγινε λόγος για την σύραξη στη Γεωργία, για την ιστορική αναδρομή, ποιος άρχισε κλπ αντικειμενικά μπορούμε να πούμε ότι ε, Ρώσοι ε, στρατιώτες ευρέθηκαν παράνομα στη Γεωργία, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Ο κύριος Μποστινάρου αναφέρθηκε σε κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί όταν υπάρχει διαφορετική ε, κατάσταση στις χώρες μας, οικονομική και γενικότερη. Είναι δύσκολο να έχουμε ενότητα ε, αλλά στην ε, πολιτική γειτονία ε, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ισχυρή και ισόρροπη και αυτό έχουμε και στη σχέση μας με τη Ρωσία με κάποιες βασικές δεσμεύσεις που διέπουν τη σχέση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Ας χειροκροτήσουμε τα μέλη του πάνελ. Κυρία, κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο και συνεισέφεραν στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μέρης της

Colleagues, I kindly ask... Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε με κάποιες πληροφορίες που έχω για εσάς. Υπάρχουν στην αίθουσα μέλη του Αφρικανικού Κοινοβουλίου οι οποίοι έχουν από καιρό ζητήσει να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μία ενημέρωση ε, της Επιτροπής, Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας για την αποστολή στην Ιταλία και τη Μεσόγειο. Έτσι ώστε να γίνει ένας απολογισμός της αποστολής τρίτων. Επισκεφθήκαμε αρκετούς οργανισμούς, κεντρικούς κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ιταλία, τοπικούς οργανισμούς, δεν πήγαμε μόνο στη Ρώμη δηλαδή και στα περίχωρα, αλλά και στη Σικελία, Κατανία. αλλά και σε επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, την επιχείρηση Σοφία και πήγαμε στην ε, Νάπολη στα γραφεία του ΝΑΤΟ. Είχαμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ήμασταν μόνο τρεις μέρες από τις 17 ως τις 19 Ιουλίου. Επικεφαλής της αποστολής ήμουν εγώ. Στη συμμετοχή, ε, στην αποστολή συμμετείχε επίση ο κύριο Κιέζα, ο Ιβο Μπελέτ από το Βέλγιο και ο κύριος Φρουντζουλίτσα από τη Ρουμανία. Επίσης, μας συνόδευσε ο Σαλβατόρ Πολιέζε, ο οποίος είναι βουλευτής ε, της ε, περιοχής εκεί, της Κατάνια και η συνεισφορά του ήταν πολύτιμη. Θεωρώ πως ήταν από τις πιο εξαντλητικές αποστολές που έχουμε κάνει, ακριβώς διότι επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, κάθε μέρα πηγαίναμε αλλού από τη Ρώμη στην Νάπολη και την Κατάνια. Νομίζω όμως πως ήταν ιδιαίτερα καλή αποστολή, ενημερωτική και ωφέλιμη. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο... Α, όχι, δεν είναι εδώ ο κύριος Κιέζα. Συγγνώμη. Τότε λοιπόν νομίζω πως θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό, να γίνει σωστά ενημέρωση έτσι ώστε να πληροφορηθούν όλα τα μέλη για το τι συνέβη. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, υπόλοιπους συμμετέχοντες, τους συνομιλητές μας, για τον ανοιχτό χαρακτήρα που έδειξαν, τον άψογο επαγγελματισμό τους και τη διάθεσή τους να μοιραστούν μαζί μας γνώση, εμπειρία και για το κλίμα συνεργασίας που έδειξαν. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με το μεταναστευτικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια λοιπόν που πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά η ενημέρωση και να είναι εδώ όλοι οι συμμετέχοντες στην αποστολή. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν ε, το χρόνο με μία αναβολή για κάποια στιγμή στο μέλλον, έτσι ώστε να ενημερωθούμε καλύτερα. Η επόμενη συνεδρίαση μας θα είναι στις 23 Σεπτεμβρίου και θα προσπαθήσουμε τότε να συμπεριλάβουμε το θέμα στην ημερησία διάταξη. Και τώρα το επόμενο σημείο είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο σχέδιο έκθεσης, ετήσιας έκθεσης για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Περιέχονται αποφάσεις συμβουλίου, πρωτοβουλίες της είπα της εκπροσώπου, αντιπροέδρου. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στον εισηγητή κύριο Γκάλερ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Με χαρά σας παρουσιάζω σήμερα το σχέδιο της έκθεσης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Είναι μοναδική η κατάσταση. Βλέπουμε να επιδεινώνεται η κατάσταση στην ασφάλειά μας μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου προς Ανατολάς και Συζητήσαμε τόση ώρα για το ρόλο της Ρωσίας στην ε, ε, Ουκρανία και τις ε, απειλές για τον κυβερνοχώρο και στις χώρες μας. Στο Νότο εγκληματίες και τρομοκράτες είναι ενεργοί και από το Σαχέλ και πέρα από τη Μεσόγειο επεκτείνεται αυτή η αστάθεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείες τελειοποιούν και οριστικοποιούν μάλλον τι ε, σχέσει του με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά ε, το Brexit. Βεβαίω είναι προσιλωμένη πλήρω η ε, Βορειοατλαντική Συμμαχία, αλλά η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ίδια με το παρελθόν. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και εκείνου. Ε, που υπηρετούν άνδρες και γυναίκες σε τρεις υπήρους, στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζουν το σεβασμό μας και τη συνεχή μας υποστήριξη, διότι είναι στην πρώτη γραμμή για να οικοδομηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια και ε, να εξασφαλιστεί η δική μας ασφάλεια των πολιτών μας. Οι μελλοντικέ δυνατότητες ε, θα πρέπει να είναι προ όφελο ε, του πληθυσμού των ανδρών και γυναικών και όχι την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Καλά, μπορεί και η βιομηχανία λίγο να υποφεληθεί, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και δυνατότητα παρέμβαση. Είναι έχει έρθει η ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση πρόσφατες δράσεις άλλων θεσμικών οργάνων δείχνουν ότι προχωρούμε και είναι ελπιδοφόρο όλα αυτά. Μετά την παρουσίαση της Παγκόσμιας Στρατηγικής πέρσι, και την έναρξη των εργασιών σε επίπεδο κρατών μελών. Έχουμε ε, κοινέ αποφάσει για την άμυνα εκτελεστικέ. Οι αντιπρόεδροι Κατάινε, ε, Μογκερίνη και η Επίτροπο Μπιακόφσκα έδειξαν πολιτικό θάρρο και όραμα τον Ιούνιο όταν παρουσίασαν την ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, νομοθετική πρόταση για ε, ένα πρόγραμμα αμυντική βιομηχανία και ένα έγγραφο προβληματισμού για την άμυνα. Τέλο, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ φαίνεται να είναι ενεργή μετά την απόφαση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε πάνω από 42 τομείς. Συμπεραίνω με χαρά ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμμετέχουν στην υλοποίηση του πολιτικού οράματος που γεννήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στη δική μας Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Για το όραμα αυτό συνεργαστήκαμε και σε προηγούμενες εκθέσεις. καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μας μιμηθούν, να μας αντιγράψουν και δεν πρόκειται να σας μηνύσουμε για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λεγοκλοπής. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και στο παρελθόν και αυτό με ενέπνευσε για τη σημερινή έκθεση. Με την έκθεση αυτή έχουμε τώρα την ευκαιρία να δώσουμε συνέχεια στην καλή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα αριθμό κρατών μελών συμφωνούν με τη μόνιμη διαφρομένη συνεργασία και την ευάθυνση στον τομέα αυτό. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνει όλο και περισσότερο τα πιο περίπλοκα ε, θέματα και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα κράτη-μέλη στη βελτίωση των στρατιωτικών του συνατοτήτων και ικανοτήτων. Ε, και είναι επίκαιρη η πρόταση για το αμυντικό ταμείο. Πέρσι δεσμευτήκαμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα και μαζί με το Συμβούλιο προχωρήσαμε σε μια προπαρασκευαστική δράση για την ε, έρευνα στην αμυντική βιομηχανία και χαίρομαι που δίνεται συνέχεια και υποστηρίζεται αυτή η προσπάθεια από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Στις 7 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε μια δική της πρόταση για συγχρηματοδότηση ανάπτυξης ε, στρατιωτικών δυνατοτήτων. Έρχεται αυτό να ε, πληρώσει ένα διαφορετικό κενό που υπήρχε για τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων για να βελτιώνουν τα κράτη-μέλη της δυνατότητές τους. Μετά τις προτάσεις αυτές, οι βουλευτές και η Επιτροπή μας παραμένουν ενεργοί, έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσουμε, πρώτα απ' όλα στη συζήτηση και τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι πρέπει να αποφασίσουμε 40 εκατομμύρια για τον προϋπολογισμό του 2018 για την έρευνα στην άμυνα. Θα πρέπει να αρχίσουμε συζητήσεις για τα 500 εκατομμύρια που υπάρχει πρόθεση να δαπανηθούν στο αμυντικό πρόγραμμα το 2019 και 2020 πάντα για την έρευνα. Εγώ προτείνω να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και να εγκρίνουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα μελλοντικά χαρακτηριστικά. Εγώ προτείνω να αναπτυχθεί η αμυντική βιομηχανία με ξεχωριστό προϋπολογισμό και δικού τους κανόνες στο επόμενο πολιτεύστημο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της αμυντικής βιομηχανίας, ε, θα πρότεινα να διευρυνθεί η νομιμότητα αναφερόμενη στο βασικό στόχο ότι στόχος είναι ε, να έχουμε μια κοινή ε, αμυντική πολιτική, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε νέους στρατηγικούς στόχους και θεσμική συνεργασία στο δρόμο προς την αμυντική ένωση. Επανέρχομαι στην έκθεσή μου, ε, όπου ζητούσα μια λευκή βίβλο για την ασφάλεια και την άμυνα καθορίζοντας παγκόσμια θέματα άμυνας, θα πρέπει όλα αυτά να είναι συνδυασμένα και όχι κατακαιρματισμένα σε ένα ενιαίο έγγραφο προς την Αμυντική Ένωση. Η Επίτροπος Βιανκόφσια και η Γενική της Διεύθυνση ε, εργάζονται πάρα πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε, να έρθουμε πιο κοντά ε, με το έργο των διαφόρων ε, Υπουργείων μείνει στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει και θα γίνει καλύτερα αν υπάρξει μια ε, Γενική Διεύθυνση Άμυνας. Αυτή μαζί με τον Ευρωπαϊκό ε, Αμυντικό Οργανισμό θα έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν ε, υποστηρικτικό προς τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Αυτά τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε η Λευκή Βίβλος να γίνει ένας μηχανισμός ετήσιος αναθεώρησης. Υπάρχει σήμερα που λέγεται CART συντονισμένος ετήσιος μηχανισμός αξιολόγησης για να δούμε πώς προχωράει η προσπάθεια στα κράτη-μέλη, στην έρευνα και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Επιπλέον τα κράτη-μέλη, ένας βελτιωμένος αμυντικό οργανισμός και η μελλοντική Γενική Διεύθυνση άμυνα, θα πρέπει να έχουν μια μόνιμη δομημένη συνεργασία που ελπίζω να στηθεί μέχρι τα τέλη του έτου. Ελπίζω να υποστηρίξετε τι προτάσει μα για να έχουμε και μια ετήσια κοινοβουλευτική έκθεση που βεβαίω έχει σημασία για του πολίτε μα. Θα πρέπει τα άλλα θεσμικά όργανα να έχουν μια καλύτερη αξιολόγηση από πλευρά μα του έργου του και να προτείνουμε νέε ιδέε για την πορεία μα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Thank um, Αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν δύο σκιώδεις στους σοσιαλιστές. Νομίζω ότι ο κ. Μποστινάρο είναι αυτός που θα πάρει το λόγο. Ναι, εγώ είμαι παρόν μόνος, θα μιλήσω όμως και για τους δύο μας. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Γκάλερ για την εξαιρετική του πρόταση. Είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης και κατά κάποιο τρόπο μπορεί έτσι η υποεπιτροπή μας να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία έχουν αρχίσει να είναι οι βασικές μας προκλήσεις αλλά θα είναι όχι απλώς βασικές, υπαρξιακές τα χαρακτήριζα, στα πλαίσια ενός ε, δραματικά θα έλεγα αλλαγμένου περιβάλλοντος στον τομέα της ασφάλειας. Θα ήθελα λοιπόν να ε, διευρύνουμε όμως λίγο περισσότερο την αναφορά μας ε, στην τρομοκρατία γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απαιτεί θα έλεγα να υπάρξουν άμεσες δράσεις και νομίζω ότι δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις. Μας ανησυχεί επίσης η πολυμορφία της τρομοκρατίας και των προκλήσεων που δημιουργεί, όπως επίσης και η εμφάνιση του λεγόμενου, της λεγόμενης τρομοκρατίας χαμηλού κόστους, low cost terrorism, βλέποντας τις τελευταίες επιθέσεις, φαίνεται ότι αυτού του είδους οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι από τις πιο δύσκολες να αντιμετωπιστούν. Κάποιες προτάσεις επίσης για την καταπολέμηση των πηγών της τρομοκρατίας, και επίσης η απορριζοσπαστικοποίηση των νέων και ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδράμει στην απορριζοσπαστικοποίηση εμπνεωμένη από τα προγράμματα τα οποία ακολουθήσαμε στη Βοσνία, Ευζεγοβίνη και στο Κωσυφοπέδιο. Θυμηθείτε πόσοι πολεμιστές ακραίοι υπήρχαν εκεί και οι οποίοι τώρα έχουν μετατραπεί θα Νομίζω επίσης ένα άλλο τομέα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Η αμοιβαία ενημέρωση είναι ένα βασικό πρόβλημα και ελπίζω να υπάρξουν προτάσεις από πλευράς των νομοθετικών οργάνων για την αντιμετώπιση των κενών και για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και με άλλους οργανισμούς σημαντικούς όπως ε, το ΝΑΤΟ και με τρίτες χώρες. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, να αναφερθώ επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τους κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΑΣΕ, Ηνωμένα Έθνη, Αφρικανική Ένωση και Αραβικό Σύνδεσμος. Και για μια ακόμη φορά έχω αναφερθεί στο ΝΑΤΟ βέβαια, σήμερα βλέποντας το πώς έχουν τα γεγονότα και όχι μόνο η ρητορική, είμαι πεπισμένη ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες εμένουν στις αξίες του ΝΑΤΟ, εμένουν στην χρησιμότητα του άρθρου 5 και το κοινό ψήφισμα το οποίο υιοθέτησε το, ε, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία για τις σχέσεις με τη Ρωσία δείχνουν ότι γενικά η καθεστική ατάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες θέλει ε, να υπερασπιστεί τις αξίες και το ρόλο του ΝΑΤΟ που ε, παραμένει υψηλή σημασία για τη συλλογική μας άμυνα. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ λίγο περισσότερες αποχρώσεις έτσι ώστε να υπάρξει αναφορά σε αυτές τις εξελίξεις. Είχαμε πάει στη ΣΥΠΑ μία εβδομάδα πριν από την υιοθέτηση του κοινού ψηφίσματος ανάμεσα στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και νομίζω ότι ήταν σαφής η βούληση και η υποχρέωση την οποία εξέφασαν και τα δύο κόμματα να προφήσουν την γραμμή του σεβασμού του ΝΑΤΟ και να υπογραμμίσουν ότι θα εξαναγκάσουν τον Τραμπ να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική. Ε, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα σας ευχαριστώ για την πρότασή σας, όχι μόνο γιατί προερχόμαι από μια χώρα η οποία πράγματι εμπλέκεται και επιθυμεί την Ευρωπαϊκή Έμεινα, αλλά να επαναλάβω εδώ δύο σημεία. Πρώτον, η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Άμυνα να καλύψει τις ανάγκες ασφαλείας και τις ανάγκες της αμυντικές όλων των κρατών μελών. Θα πρέπει να είναι τμήμα της απάντησής μας στα προβλήματα ασφαλείας. Και δεύτερον θα ήθελα να μετριάσω τον ενθουσιασμό κάποιων ότι η άμυνα της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζεται στη βασική αρχή αγορά στα ευρωπαϊκά προϊόντα και όπλα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, μια τέτοια λογική μπορεί να βοηθήσει και να λειτουργήσει ενοποιητικά. Αν όμως εμείνουμε σε κάποιες άλλες ε, ε, πλευρές οι οποίες δυστυχώς δεν μας βρίσκουν σύμφωνος, τότε θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Να βάλουμε περισσότερες αποχρώσεις και νομίζω ότι οι εξελίξεις και τα δημοσιονομικά για την κάλυψη των αναγκών για το Ταμείο Άμυνα στο μέλλον έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ίδια την ύπαρξη της Ένωσης. Και να αναφερθώ εδώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μακρόν έχουμε να, κάνει μια, να κάνουμε με μια Ευρώπη η οποία είναι σε θέση να προστατεύει και να αμήνεται. Σωστά. Αλλά αυτό πρέπει ε, να μην μείνει στα λόγια, να γίνει πράξη. Το να πούμε ότι είμαστε υπέρ της άμενας της Ευρώπης ε, δεν σημαίνει τίποτα. Να θυμίσω εδώ ε, κάτι το οποίο έλεγε ένας Αμερικανός στρατιωτικός στο Συμβούλιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συνειδητοποιείτε τι σημαίνει να είστε μέλος του ΝΑΤΟ. Σημαίνει ότι πρέπει να είστε έτοιμοι να κάνετε πόλεμο, όχι να μιλάτε για πόλεμο, αλλά να πολεμήσετε και να κερδίσετε τον πόλεμο. Εμείς λοιπόν θα πρέπει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Άμυνας να προστατεύσουμε τις ανάγκες ασφαλείας μας όχι μόνο επιμέρους Προφανώς όχι πλήρως και απολύτως γιατί αυτό τεχνικά, πολιτικά και στρατηγικά δεν είναι εφικτό αλλά η ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να είναι τμήμα της συλλογική μας άμυνας ε, συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με το ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μποστινάρου για την ομάδα ΕΣΥΑΡΟ. Ο Τζέφρι Βανόρδεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον ε, Μιχαήλ Γκάλερ και την έκθεσή του σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του κινδύνου, την εκτίμηση της απειλής και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η στήριξή μου τελειώνει εκεί. Διότι ο Μίχαελ επιχειρηματολογεί, και δεν το λες κιόλας Μίχαελ, επιχειρηματολογεί υπέρ μιας ε, Ευρώπης ε, συγκεντρωτικής επιπέρ ενός ευρωπαϊκού στρατού. Και συμφωνώ και με τα όσα είπε ο κύριος Μποστινάρου. Πολλά λέγονται, ουσία καμία. Αποτελέσματα μηδέν. Δεν ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως είναι ο μόνος και και θεματοφύλακας των δυτικών αξιών και ο μόνος που έχει δικαίωμα και δυνατότητα να προστατεύει τα συμφέροντα και τις αξίες αυτές. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είπατε πως ε, επανεκτιμούν τη θέση τους απέναντι στο ΝΑΤΟ. Όχι, καθόλου, καμία σχέση. Και η μία χώρα και η άλλη ζητά ένα ενισχυμένο ΝΑΤΟ. Εάν ε, το λέτε εσείς αυτό νέο ναι, ορισμό, εντάξει, αλλά σε καμία περίπτωση οι Ηνωμένε Πολιτείε ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουν να επανακαθορίσουν τη σχέση τους με το ΝΑΤΟ. Όχι, όχι, δεν, μην προσπαθείτε να ξεγλιστρήσετε. Είπατε ΝΑΤΟ, είπατε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύει αυτό, Μίχαλ, και πρέπει να αλλάξει στο κείμενο. Μετά, στην παράγραφο 30. Θε να δημιουργηθεί μια γενική διεύθυνση άμενα μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην ουσία ίσως αυτό που θα ήθελες είναι ένα Υπουργείο Άμυνα για την ευρωπαϊκή σου κυβέρνηση. Και ακριβώς όπως ε, το είπες, αυτό θα είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν. Και αναρωτιέμαι τι θα πούν τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Αν ρωτούσαμε τους πολίτες των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, εάν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τις εναποθέτουν την ε, ασφάλειά τους, τότε η απάντηση θα ήταν αρνητική, μηδενική εμπιστοσύνη. Μετά αναφέρθηκε στις αποστολές στα πλαίσια της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αλλά δεν νομίζω πως ε, αυτοί που συμμετέχουν στι αποστολές θεωρούν πως υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στρατιωτικό προσωπικό που έχει πάει να κάνει ε, κάποια στρατιωτική δουλειά. Πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Και δεν νομίζω πως θεωρούν ότι αυτά που κάνουν είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν εδώ τα πράγματα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση ως επιλώνας του ΝΑΤΟ νομίζω είναι μια πρόταση που αγνοεί το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία είναι οι δύο πολύ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ οι οποίες ε, στα επόμενα χρόνια δεν θα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία τουλάχιστον. Αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή φυσικά είναι το Brexit. Και υπάρχει μία ελάχιστη αναφορά σε αυτό κάπου, δεν θυμάμαι πού το είδα. Αναφέρεται ότι, α ναι, και θέλουμε και νέα, νέα έδρα για την ε, ΝΑΦΟΡ. Ναι, όμως, εφόσον μιλάμε για την πολιτική ασφάλειας και άμυνα στην Ευρώπη, πρέπει να αναγνωρίσουμε το ότι η πιο ισχυρή στρατιωτικά δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, αποχωρεί και νομίζω πως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε ποιο θα είναι το μέλλον των σχέσεων της Ένωσης με τη χώρα αυτή. Αφήστε τον ΝΑΤΟ κατά μέρου. Οι μελλοντικέ σχέσεις της Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο Ποιε θα είναι και μπορώ αν θέλετε να σας ε, κάνω και συγκεκριμένη διατύπωση των ε, προτασεών μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ζωράντος εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλερ. για την εξαιρετικά ποιοτική έκθεσή του. Η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας τώρα βρίσκεται σε στάδιο αλλαγής και ενδεχομένως υπάρξει και πρόοδος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ λογικό η ετήσια έκθεση να εστιάζει στις αλλαγές αυτές. Όμως, έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της αμυντικής πολιτικής, του Ταμείου Άμυνας, του Ταμείου αμυντικής έρευνας και του προγράμματος ε, της ε, άμυνας και της βιομηχανίας. Όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει δρομολογηθεί. Ορισμένα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης αυτή τη στιγμή κάνουν μόνο δηλώσεις. Πρώτα πρέπει να δούμε αποτελέσματα αυτής της νέας πολιτικής άμυνας. Γι' αυτό και θα στηρίξω απόλυτα το σχέδιο έκθεσης και τη θέση του σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Τον προϋπολογισμό στο διεθνές, στο, διεθνές... Ε, στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τη χρηματοδότηση και τις task force που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της συνεργασίας. Φυσικά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και νομίζω πως πρέπει να είμαστε σαφέστεροι σε ό,τι αφορά το μόνιμο στρατηγείο και εκ μέρους των θα θέλαμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες και να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση θα πρέπει να γίνει ένας ε, γνήσιος πυλώνας του ΝΑΤΟ, κάτι που δεν είναι και είναι κάτι που λείπει. Και είναι μια ευκαιρία 17 χρόνια μετά την ε, δημιουργία της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας να γίνει πρόοδος. έτσι ώστε να πάμε σε μια πραγματική αμυντική πολιτική και σε μια αληθινή αμυντική ένωση. Πολλά εμπόδισαν την πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όμως εμείς έχουμε τη δυνατότητα διαμόρφωσης της πολιτικής αυτής. Σίγουρα είναι απαιτητικό το έργο μας, όμως πρέπει να δράσουμε. Του χρόνου θα έχουμε την αναθεώρηση των δυνατοτήτων και εκεί θα φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες και εάν έχει τη δύναμη να προοδεύσει πραγματικά και να προχωρήσει την πολιτική άμυνας εάν μπορεί να χειριστεί τα όπλα, τα οπλικά της συστήματα και να διαχειριστεί και μερικά πολύ βασικά ζητήματα άμυνας τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Θα δοκιμαστεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις προκλήσεις αυτές ε, τόσο στη γειτονία της όσο και από τις απειλές που δέχεται. Εδώ λοιπόν πρέπει να δείξουμε τη δύναμη για να γίνει πραγματική πρόοδος. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Λόζινγκ, εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ο κύριος Βαν Όρντεν, θα αρχίσω από τα θετικά. Διευκολύνει πολύ τη δουλειά μας αυτό όταν δεν έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Πράγμα που ισχύει και με την παρούσα έκθεση. Δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη. Άρα αυτό είναι θετικό. Αυτά όμως ήταν τα θετικά. Τελειώσαμε από πλευράς μας. Για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μποστινάρου, να πω ξεκάθαρα ότι εγώ δεν είμαι εδώ επειδή είμαι πρόθυμη να ε, πάω να πολεμήσω αλλά είμαι εδώ γιατί θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω τον πόλεμο. Διαβάζοντας την έκθεσή σας κύριε Γκάλερ, έχει την αίσθηση ότι είμαστε κατά μεσή στον πόλεμο όπου μας έχουν επιτεθεί διάφοροι ε, πιθανοί και απίθανοι, σαν να είναι ο Πούτιν ε, ε, έξω από τις Βρυξέλλες πρώτων τυχών, ότι μας επιτίθενται οι πάντες και θα πρέπει να αποσοφηθούν αυτές οι επιθέσεις και να παταχθούν. Δεν λέτε όμως στην έκθεσή σας τι γίνεται με τις αιτίε, για ποιο λόγο και ποιες είναι οι άνευ προηγουμένων προκλήσεις, ε, ποιες αλλαγές έχουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η προοπτική να αλλάξει, να δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε τις Αιτίε τη επιδείνωση αυτής τη εξωτερικής πολιτικής για να είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Καλωσορίζεται ρητά μεταξύ άλλων ε, στις παραγράφους 5, 11 και 22 τις διάφορες προτάσεις των τελευταίων μηνών. Το Αμυντικό Ταμείο, μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, ΠΕΣΚΟ, ε, στρατηγείο κτλ έχω την εντύπωση ότι έχουμε τώρα ένα κίτ εδώ για να... Ε, μάλλον ένα, ένα είδος, ε, πώς να το πω, ε, συγκολητικής για να ενώσουμε τα διάφορα κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σπάσει. Η κυρία Μογκερίνη είπε ότι τους τελευταίους δέκα μήνες πετύχαμε περισσότερα από ότι την τελευταία δεκαετία. Οι περισσότεροι αυτό θα το θεωρήσουν πολύ καλό, αλλά εγώ προσωπικά και η πολιτική μου ομάδα έχουμε θορυβηθεί βαθύτατα. Επειδή λοιπόν δεν είναι έκπληξη η έκθεσή σας, δεν θα σας εκπλήξει και η στάση της δικής μας πολιτικής ομάδας. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για σας, γιατί δεν σας εκπλήσει ότι ε, απορρίπτουμε την Αμυντική Ένωση και τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν πιστεύουμε ότι έτσι βελτιώνεται σημαντικά η ασφάλεια των Ευρωπαίων. Βελτιώνεται η οικονομική ασφάλεια της αμυντικής βιομηχανίας από την άλλη. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στο άρθρο 41.2 της Συνθήκης Λισαβόνας απαγορεύονται ε, να χρηματοδοτούνται τέτοιες στρατιωτικές δράσεις από τον Ευρωπαϊκό ε, ε, Προϋπολογισμό. Τώρα ορισμένοι αποπειρώνται να τα μεταθέσουν όλα αυτά στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Είπατε κύριε Γκάλερ ξεκάθαρα και καλά κάνατε τις προθέσεις σας δηλώσατε ότι θέλετε προοδευτικά να προχωρήσετε προς μια κοινή αμυντική πολιτική. Τουλάχιστον ξέρουμε που το πάτε, στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Δηλαδή εκεί υπάγεται αυτό και όχι στην ε, αμυντική ε, πολιτική, μάλλον στην βιομηχανική πολιτική, οπότε απαγορεύεται η χρηματοδότηση. Μια κούρσα εξοπλισμών θέλετε, απλούστατα. Εμείς αποκρύουμε οποιαδήποτε απόπειρα ε, χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό να χρησιμοποιηθούν προς αυτό το σκοπό για αμυντική έρευνα. Μιλάτε και για Γενική Διεύθυνση Άμυνας ε, στις παραγράφους 13-15 και συνεργασία με ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Διαφωνούμε και σε αυτό και ζητούμε έντονα να γίνονται σεβαστά τα κοινοβουλευτικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου και να ενισχυθούν απέναντι στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό. Τώρα θέλετε Γενική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά για την άμυνα. Αυτό θα ενίσχυε τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήταν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Τώρα δεν πρόκειται να σας πω ε, άλλες λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω. Σύντομα, συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, στόχος αμυντικών δαπανών 2%. Πιστεύω ότι οι πολίτες στα κράτη-μέλη διαφωνούν, τουλάχιστον στη Γερμανία δεν το επιθυμούν οι πολίτες. Ρίζω δημοσκοπήσεις που το ε, διαψεύδουν αυτό. Ο κόσμος διαφωνεί. Δεν θα σας εκπλήξει τελικά ότι δεν θα υπερψηφίσουμε την έκθεσή σας και θα κάνουμε και τροπολογίες αλλά και έκθεση μειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαλέρο, με τον Πρασίνων. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ όταν διάβασα την έκθεση αυτή έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία δεν μπορώ να στηρίξω. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που κρίνω υπερβολικές. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτά με τα οποία συμφωνώ. Καταρχάς είμαστε υπέρ του να πούμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Έχει αλλάξει και η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι λοιπόν θετικό να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία, μια βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες χώρες μέλη. Πιστεύουμε επίσης ότι τίθενται και το θέμα της ανάγκης επενδύσεων στην πολιτική άμυνας και στην αμυντική βιομηχανία, αλλά πέραν αυτού όχι. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τίθενται στην έκθεσή σας με τα οποία διαφωνούμε. Γι' αυτό και θα, θα καταθέσουμε τροπολογίες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι βασικό για μας έχει σχέση με την οικονομία. Ε, υψηλότερος προϋπολογισμός λοιπόν στις στρατιωτικές δαπάνες δεν μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι στα κράτη-μέλη έχουμε έναν προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες ιδιαίτερα σημαντικό. Και αν πράγματι θέλουμε να συνεργαστούμε, ας εξοικονομήσουμε χρήματα και όχι να δαπανίσουμε περισσότερα που θα αφαιρεθούν από τα κοινωνικά ταμεία, από τα διαφορετικά συγγνώμη ταμεία μπορούμε να συνεργαστούμε με καλύτερο τρόπο όχι μόνο στον τομέα της άμυνας και όχι μόνο στον τομέα των δημοσιονομικών αλλά είμαστε κατά των προτάσεων για αύξηση των δαπανών σε άλλους τομείς. Και θα καταπολεμήσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος στο Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες διαφωνούν δεν ε, προκαταλαμβάνω τις θέσεις άλλων χωρών, εγώ αναφέρομαι στη δική μου. Λοιπόν, ε, ίσως στην έκθεσή σας λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πραγματικής ε, επιρροής της οικονομίας, να στηριχθούμε σε αυτά τα οποία κάνουμε και να τα βελτιώσουμε. Μία ακόμα παρατήρηση γίνεται αναφορά ε, πολύ συνοπτική στην Βόρεια Κορέα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι κάπως πιο αναλυτική. Έχουμε μια πολιτική μη διάδοση των πυρηνικών όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επέμβουμε ε, με πιο ισχυρό τρόπο. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Βαν για το τι μπορεί να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που θα κατατεθεί από πλευράς μας προς την κατεύθυνση αυτή. Ενημερώνοντάς σας κυρία Βαλεά, είχαμε μια συνάντηση για την πιθανότητα στο Στρασβούργο μια συνάντηση ειδική για τη Βόρεια Κορέα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, όχι μόνο για την έκθεση, νομίζω ότι είναι επίγον να το συζητήσουμε. Και υπάρχουν και άλλα θέματα επίσης στον τομέα του αφοπλισμού. Υπάρχει εκπρόσωπος και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που θέλει το λόγο. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω ε, στις ερωτήσεις σας, αν έχετε. Ναι, ο κύριος Γκάλερ, νομίζω... Όχι, κύριε Γκάλερ, νομίζω πως δεν έχει ζητήσει άλλο συνάδελφο το λόγο. Εσείς? Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, για την αντίδρασή σας. Οι αντιδράσεις τα μάλιστα ήταν οι αναμενόμενες, θα έλεγα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα. Ο συνάδελφος κύριος Μποστινάρου Μα είπε πως ε, θα ήθελε να δει μια αναφορά στην τρομοκρατία. Θεωρώ πως ε, σε αυτήν την έκθεση πρέπει να σταθούμε στην εξωτερική διάσταση. η οποία αφορά κυρίως τομείς που σχετίζονται με τις ε, δομές στο νότο και στα νοτιοανατολικά. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το δίπολο εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια. Τώρα, αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και εδώ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν νομίζω πως ε, μπορούμε να επιβάλλουμε θεσμικά στα κρατημέλη να συμμετέχουν στις ε, επιτροπές αυτές. Αυτό δεν είναι... Ε, αυτός δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών. Θα έπρεπε όμως να τους δώσουμε μία δυνατότητα για συνάντηση και ανταλλαγή πληροφοριών εφόσον το επιθυμούν και εφόσον μπορούν. Δεν πρέπει λοιπόν ε, να προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Συμφωνώ πάντως με αυτά που είπατε. Τώρα, οι προσπάθειες άμυνας πρέπει να είναι συμπληρωματικές στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εάν ήμουν Αμερικάνος και κοιτούσα προς την Ευρώπη θα έβλεπα ένα κολάζ αμυντικό ε, πολιτικών και αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, μετά από πολλά χρόνια ε, βελτίωσης ε, της διαλειτουργικότητας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να χτίσουμε και να δώσουμε προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερα για παράδειγμα στον τομέα της πιστοποίησης θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την κατάσταση, να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Ε, γιατί τώρα ακολουθούμε περίπλοκες διαδικασίες που καθυστερούν πάρα πολύ. Πρέπει να βελτιωθούμε και να γίνουμε και πιο ελκυστικοί για τους ε, Αμερικανούς εταίρους μας. Και το Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά δεν είναι μόνο του, δεν είναι τόσο καλό που δεν χρειάζεται άλλον. Όχι, πρέπει να συνεργαστούμε. Η συνεργασία βοηθά στο να γίνεις καλύτερος. Και η ε, ΠΕΣΚΟ δεν ε, είναι ένα, μια λύση για τα πάντα, δεν είναι all inclusive θέρετρο, πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας έτσι ώστε να αυξήσουμε και την αποτελεσματικότητά μας για να γίνουμε καλύτεροι μαζί από ότι ο καθένας μόνος του. Αυτό είναι το δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε, γιατί μόνο έτσι θα γίνουμε ελκυστικός εταίρος για τους Αμερικανούς, όχι μόνο για τον ε, Τραμπ. Από την εποχή Κλίντον μας λένε πώς ε, πρέπει να συνεισφέρουμε στον ε, τομέα της άμυνας. Και τώρα η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και πρέπει επιτέλους να δράξουμε την ευκαιρία για να εντείνουμε τις προσπάθειες βελτίωσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Τώρα, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας όπως... Ε, ε, είπατε, δεν είναι ένας οργανισμός της Κομισιόν, αλλά είναι ένας οργανισμός του Συμβουλίου. Γι' αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον το προσωπικό του θα έπρεπε να πληρώνεται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και αυτός ο προϋπολογισμός να αυξηθεί κάπως έτσι ώστε να καλύψει τις ε, ανάγκες του προσωπικού. Βέβαια αυτό δεν μπορούσε να γίνει για πάρα πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, λόγω πληθωρισμού, λόγω πολλών ε, λόγων. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε, γι' αυτό λοιπόν και θα ήθελα να το αναπτύξω σε πολλές ε, παραγράφους. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε δηλαδή την ευρωπαϊκή άμυνα, πώς μπορούμε να καταρρύψουμε τα εμπόδια και τους φραγμούς που δημιουργούνται μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Ε, θα έπρεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει αντί να μπλοκάρει τα πράγματα. Γιατί νομίζω πως τα συμφέροντά μας είναι κοινά στο, στο μης αυτούς. Εμείς, ναι, ναι, εμείς αποφασίζουμε και μετά εσείς θα μπορείτε να πείτε εάν μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό το πλαίσιο ή όχι. Και μετά, κατά περίπτωση, θα καλωσορίζουμε μέλη. Όμως οι αποφάσεις ε, θα είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των μελών. Τώρα, απαγόρευση της χρηματοδότησης. Ε, μας είπατε, ε, κυρία Λόζιν, ότι υπάρχει στη συνθήκη. Ναι, έχετε δίκιο. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όμως τα ερευνητικά προγράμματα είναι διαφορετική περίπτωση. Εκεί υπάρχει μια κοινή κατανόηση ε, ότι ναι μεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά προγράμματα από τον ε, κοινωνικό προπολογισμό, αλλά όχι ας πούμε ε, μη επανδρομένα οχήματα, όχι πύραυλοι. Ή άρματα. Υπάρχει λοιπόν κάποια συνεννόηση για αυτό το θέμα, αλλά πράγματι δεν χρηματοδοτεί ο κοινοτικό προπολογισμό στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά θα χαρώ πολύ για τις τροπολογίες σας και θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού να τις ε, λάβω υπόψη. Αλλά, όπως είπατε και εσείς, ε, παραθέσατε τα λόγια της κυρίας Μογκερίνη ε, και με χαροποίησε πάρα πολύ αυτό προσπάθησα εδώ και πολλά χρόνια στην Επιτροπή με εσάς τους συναδέλφους να ε, δουλέψω. Εργάστηκα σκληρά και ευτυχώς τώρα νομίζω πως βλέπω αποτελέσματα. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο σχόλιο. Μας είπατε πως πρέπει να γίνει αναφορά σε επιμέρους ζητήματα όπως ε, για παράδειγμα Βόρεια Κορέα. Εδώ νομίζω πως ε, χρειάζεται άλλη έκθεση Υπάρχει σχετική αρμόδια έκθεση. Εδώ ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Σε αυτή την έκθεση δεν γίνεται μία γενικότερη αξιολόγηση των κρίσεων στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ε, να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας στην έκθεση Μακάλιστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών 13 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. δεύτερη συζήτηση στην Επιτροπή μας, 11 ή 12 Οκτωβρίου, μία από τις δύο μέρες, εξαρτάται από την ημερήσια διάταξη. Αλλά σε εκείνη τη συνεδρία θα το συζητήσουμε και μετά θα ψηφίσουμε στις 10 Νοεμβρίου. Α, όχι, στην Επιτροπή Εξωτερικών. Και στις 14 Δεκεμβρίου, αν δεν απατώμε, ενδεχομένως στην Ολομέλεια. Έγκριση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεδρίαση αυτή. Στα διάφορα έχουμε τίποτα. Θέλει κανεί το λόγο. Όχι. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνεδρίαση. Θυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει η χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Ευχαριστώ και όλους τους διερμηνείς. Ήταν πολύ δύσκολη σήμερα η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε και εμείς.